everyone and uh, welcome back. We have a very heavy season. Γεια σας. Σα καλωσορίζω. Είναι δύσκολο και φορτωμένο το πρόγραμμά μα, αλλά παρόλα αυτά εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο μας. Λοιπόν, μετά από αίτημα του, της ομάδας e θα δούμε πρώτα-πρώτα τα θέματα 10, 11 και 12. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξη με αυτή την τροποποίηση. Να σας κάνω και κάποιες ανακοινώσει. Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε προ το τέλο τη θητεία, οι συντονιστέ αποφάσισαν να ανοίξουν την προθεσμία υποβολή ε, ε, τροπολογιών σε μια σειρά από προτάσεις τη Κομισιόν. Γι' αυτό δεν θα οριστεί η συγητή ε, στην ΕΝΒΗ και δεν θα, οριστεί, δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση για αυτά τα θέματα σε αυτού του φακέλου όλες μαζί οι τροπολογίες θα ε, συγχωνευτούν σε μια γνωμοδότηση και θα υποβληθεί από μένα ε, ως ε, ε, από, από, εμένα ως εκ μέρους της Προέδρου δηλαδή. τα θέματα και το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Συγκριτικοί δείκτες για τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα 19 και 20 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ. Τώρα για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη η προθεσμια αποβολη υποβολή ε, τροπολογιών είναι 9η Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην ΕΝΒ θα γίνει στι 8 Νοεμβρίου. Όσον αφορά την συνδιάσκεψη των πρέσβεων, όπω γνωρίζετε κάθε χρόνο διοργανώνεται μια τέτοια συνδιάσκεψη με του ε, πρέσβει τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η φετινή συνδιάσκεψη θα γίνει στι 4 Σεπτεμβρίου την Τρίτη το απόγευμα. Και ένα από τα τρία θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η κλιματική αλλαγή. Το σχέδιο τη ημερήσιας διάταξη σα έχει αποσταλεί και σας προσκαλώ όλους να συμμετάσχετε στην ε, συνδιάσκεψη αυτή. Μετά, στις 12 Νοεμβρίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής μας στην, στο Στρασβούργο από τις 7 έως τις 9 το βράδυ για να γίνει ψηφοφορία για κάποιες επίγουσες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Θα λάβετε το σχέδιο μερικές διάταξης ε, εν ευθέτω χρόνο. Διερμηνία έχουμε σήμερα σε 20 γλώσσες και ως συνήθως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Επίσης, σας έχουν αποσταλεί συστάσεις των συντονιστών της 10ης ε, Ιουλίου και αν δεν υπάρχουν αντερήσεις θεωρείται ότι εγκρίνονται. Επίσης, Έχετε λάβει τα πρακτικά των συνεδριάσεων μας 25-26 Απριλίου, 16-17 Μαΐου και 7 Ιουνίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις έως το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Και όπως συμφωνήσαμε θα ξεκινήσουμε σήμερα με, τα σημεία, με το σημείο 10 Συντάκτηρα της γνωμοδότησης είναι η κυρία Μελά που την αντικαθιστά η κυρία Τροσινόφσκη σήμερα. Το θέμα είναι η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Κυρία Τροσινόφσκη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχωρέσετε την κυρία Μελά, η οποία δεν μπορεί σήμερα να σας παρουσιάσει αυτή την έκθεση, αλλά για λόγους οικογενειακούς χρειάστηκε να μείνει δίπλα στην οικογένειά της και σας ζητάει να τη συγχωρήσετε. Αυτό το τρίτο κείμενο της Επιτροπής ε, για τον βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων ε, ε, αναφέρεται σε πέντε παράγοντες καρκινογένους. Έχουμε τις παρατηρήσεις των διαφόρων ομάδων στις ανταλλαγές απόψεων και τροπολογίες στην Επιτροπή Έμβη για γνωμοδότηση, για την οποία ήταν συγγήτρια, και στην Επιτροπή ΕΜΠΛ για την ουσία. Γι' αυτό χρειάστηκε να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία την οποία οφείλουμε στους εργαζόμενους, την ικανότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργοδοτών και των επιχειρήσεων, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ικανότητες της δημοσιονομικές των διαφόρων εθνικών συστημάτων για την αποζημίωση των ε, εργαζομένων που εκτίθενται στις παράγοντες αυτού. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ομοιογένεια των ε, ορίων και ότι κάθε χώρα χρειάζεται να κάνει προσαρμογή μόνο για μία ή δύο ουσίες το μέγιστον. Γι' αυτό η εναρμόνιση δεν θα πρέπει να έχει μεγάλες επιπτώσεις πάνω στα διάφορα κυκλώματα. Γι' αυτό έχω μία γνωμοδότηση χωρίς τροπολογίες σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Η κυρία Μελά ελπίζει ότι θα μπορέσετε να δεχθείτε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Κάμπος, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος να ξεκινά κάποιος την παρέμβασή του με τέτοιες δηλώσεις. Ε, ε, είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι για το θέμα το οποίο μας τίθεται Στη Νότια Καταλωνία, στην περιοχή του Φλής, εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε με ευρωπαϊκά κονδύλια να ε, προχωρήσουμε στην απορρίπανση κάποιων βιομηχανικών εκτάσεων και τις συνέπειες που υπάρχουν για τον πληθυσμό, επειδή ακριβώς υπάρχουν ε, βαρέα μέταλλα και ε, οργανο ε, ουσίες ε, ε, και σε πέντε χρόνια θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και από εργασιακή πλευρά αλλά και για θέματα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος και γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε μια έκθεση για το θέμα αυτό και χαιρούμε θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή η έκθεση τον Απρίλιο στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Και για να ολοκληρώσω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα της προστασίας των εργαζομένων κατά των σχετικών κινδύνων ε, με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και επίσης θεωρώ ότι ούτε εμείς ως νομοθέτες, ούτε από τον επιστημονικό κλάδο δεν έχουμε δει και τις ψυχικές νόσους οι οποίες σχετίζονται με το θέμα τη εργασία. Ε, αναφερόμαστε σε άγχος, κατάθλιψη, ασθένειες οι οποίε ε, ε, το 2013 η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή εκτίμησε ότι ε, φτάνουν στο 1 δις στην σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν πόροι στην έρευνα και στην ανάπτυξη για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε όλους τους τομείς και αυτό σημαίνει ότι για εκατομμύρια Ευρωπαίους είναι ζωτική σημασία στο θέμα αυτό. Ελπίζω να ήμουν όντως σύντομος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Από τους σοσιαλιστές δεν έχουμε κανένα. Η κυρία Μπισνιεύσκα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στο χώρο της εργασίας μας λέει ότι το 25% των θανάτων οφείλονται ε, σε καρκίνους και νεοπλασίες. Επίσης, ε, όσον αφορά την επαγγελματική έκθεση, το κόστος είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν στόχο έχουν να ενισχύσουν το επίπεδο προστασίας και οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θα πρέπει να είναι οι προτάσει που θα υποστηρίξουμε, διότι οι κατάλληλε συνθήκε εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικέ για αυτού οι οποίοι ε, εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει παρουσία καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων. Ε, πρέπει να υπάρχουν τιμέ αναφορά ε, για πέντε ουσίε, οι οποίε είναι καρκινογόνες και σίγουρα αυτό θα βελτιώσει την ε, ποιότητα ζωής των εργαζομένων και κατά συνέπεια θα μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερες συνθήκες εργασίας ε, στην Ευρώπη. Ε, ώστε να αποφεύγουν και επώδυνες ε, θεραπείες ε, και διάφορα προβλήματα τα οποία είναι συναφή με τον καρκίνο. Ε, ε, πιστεύω ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, αλλά αν εξετάσει κανείς τις αλλαγές που προτείνονται στο παράρτημα στην οδηγία 2004-37, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα υποβάλω λοιπόν κάποιες τεχνικές τροπολογίες, διότι χρειαζόμαστε κάποιες μικροαλλαγές. Θεωρώ ότι μια σημαντική αλλαγή θα είναι η αλλαγή που αφορά τα μέταλλα και τις ανόργανες ουσίες. Υπάρχουν συλλογικές τιμές για τις τιμές έκθεσης ε, ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να είναι ξεχωριστή κάθε τιμή και επίσης θεωρώ ότι οι τιμές αναφοράς για το κάδμιο και ο χρόνος ε, μύθιας ζωής είναι πολύ σύντομος, θα πρέπει να είναι στα 10 χρόνια. Ε, θα ε, υποβάλλω λοιπόν κάποιες τροπολογίες ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και να μην είναι αμφίσιμες οι ερμηνείες. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από τους φιλελευθέρους που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Από την ΚΟΥ, από τους Πρασίνους. Ωραία λοιπόν. Δεν έχουμε εδώ άλλους και οδηστάκτες να δώσω το λόγο στους υπολείπους. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Αν όχι, να δώσουμε το λόγο στην κυρία... Α, συγγνώμη. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορώ να παρακολουθήσω τη συζήτηση για αυτή τη ε, σημαντική πρόταση για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους ε, παραγόντες. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπο, η κυρία Τάισεν ε, δραστηριοποιείται πολύ στον τομέα, διότι ο καρκίνο ε, είναι η βασική αιτία θανάτου στον χώρο τη εργασία και ξέρουμε ότι ο επαγγελματικό καρκίνο είναι κάτι που είναι αντιμετωπίσιμο και λαμβάνονται μέτρα και η πρόταση αυτή, όπω και οι προηγούμενε, αναπτύχθηκαν σε σημαντική συνεργασία με του κοινωνικού εταίρους. Θα θέλαμε να ακούσουμε τι αλλαγέ που θα προτείνει η Επιτροπή σα κυρίω ε, όσον αφορά την ακρίβεια και τις αλλαγές για το κάδμιο και εκ παραλλήλου στην πρόταση αυτή ε, συζητιέται και στην Ομάδα Εργασίας Κοινωνικών Θεμάτων στο Συμβούλιο και εκεί θεωρούμε ότι υπάρχει αντίστοιχα επικοδομητική συζήτηση. Ο, κοινώνα, ο των κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Κοπενχάγη και πιστεύουμε ότι υπάρχει δικαίωμα των εργαζομένων να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και θα πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. Θα περιμένουμε λοιπόν την έκθεσή σας και από εκεί και πέρα θα απαντήσουμε κι εμείς. Είχα μια πιο μακροσκελή δήλωση, αλλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος ε, δεν ε, θα σας πω περισσότερα. Υπάρχει αξιολόγηση επιπτώσεων, είναι 168 σελίδες, τις οποίες αναφέρονται όλες οι οριακές τιμές ε, και επίσης και τις συνέπειες αν έχουμε υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές, οι οποίες υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη. Εξετάζονται λοιπόν και εναλλακτικέ ε, λύσει στι ε, προτάσει που έχουμε κάνει εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόταση ω έχει αυτή τη στιγμή στηρίζεται και από του κοινωνικού εταίρου και από την ομάδα εργασία ε, για την ασφάλεια τη εργασία και υποστηρίζεται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών και θεωρούμε ότι έχουμε μια εύρωστη πρόταση και θέλουμε να ακούσουμε και τις απόψεις σας και να διαβάσουμε και τη συμβολή σας στην έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρουσένσκη στη συνέχεια. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, κυρία Πρόεδρε. Απλώς θα διαβιβάσω όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων στην κυρία Μέλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, ε, στις, την 1η Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Τώρα περνάμε στην, ε, στο 11, στα, δύο θέματα, 11 και 10, σχετικά με μια, με μια συμφωνία εταιρική. Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. And, uh, uh Επίσης ε, είναι ένα θέμα ε, με το οποίο ασχολήθηκε η κυρία ε, μελά για, μια, για ένα σχέδιο χρονομοδότησης και πάλι δίνω τον λόγο στην κυρία Τροσίνσκι για να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να επανέλθουμε στο σχέδιο, η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας είναι η μεγαλύτερη εμπορική ένωση που σύναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ε, καλύπτει πάνω από το 1 τρίτο του ε, παγκόσμιου ε, ΑΕΠ και θα μπορούν τα γεωργικά προϊόντα να εισέρχονται αδασμολόγητα στην Ιαπωνία και της ε, αρχή λειτουργίας. Χάσαμε την ευκαιρία τότε, χάσαμε την ευκαιρία στον ΠΟΕ, χάνουμε τώρα και την ευκαιρία με την Ιαπωνία. Θα έλεγε κανείς ότι τουλάχιστον τώρα που ήμασταν οι δυο μας, Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία, θα μπορούσαμε να, να το είχαμε αξιοποιήσει αυτή την κοινή αρχή. Τη χάσαμε την ευκαιρία. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η αύξηση των εμπορικών συνολόγων, χωρί να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από άλλα ζητήματα όπω είναι το περιβάλλον και απλά ε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση η οποία λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κτλ. Ναι, βεβαίω. Όμω αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να υλοποιούνται στην πράξη. Όσο δεν γίνεται αυτό, εμεί δεν μπορούμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μα σε αυτά τα κείμενα που μα υποβάλλεται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εκχότ, λέει πρόεδρο. So, good to have you back. Um, we still have uh, one of the shadows, Mr. Omar G κύριος Μαματζή, Σκιώδης. Κυρία... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, από τις θερινές διακοπές, ξεκούραστοι, χαρούμενοι που ξαναβρισκόμαστε. Αλλά ήδη οι εκθέσεις που μας προτείνονται μας κάνουν κακό Και όπως είπε συνάδελφος, βρίσκεται φυσικό σε μια δημοκρατία που λειτουργεί κανονικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακάμπτεται με αυτό το σημείο. Η δημοκρατία να δέχεται τέτοια επίθεση. Όταν είδαμε τον πρόεδρο Γιούγκερ στις 17 Ιουλίου να υπογράφει αυτή την συμφωνία χωρίς καμιά στιγμή προηγουμένως να έχει ε, λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέμε, μα αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί αυτό να διαρκέσει. Το ίδιο έγινε για το ΤΑΦΤΑ, για τη ΣΕΤΑ και συνεχίζοντας έτσι η απόρριψη των ευρωπαϊκών θεσμών θα βαίνει αυξανόμενη εφόσον η συμφωνία αυτή ε, είναι η, συμφωνία που αφορά όλο και περισσότερο ε, το περιβάλλον και έχουμε έλλειψη εδώ ε, συνέπειας μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών. Είναι τελείως σχιζοφρενής από τη μία πλευρά. Είμαστε στις διασκέψεις των μερών, θέλουμε τις καλύτερες προθεσμίες για να προχωρούμε για τα διάφορα πρωτόκολλα και στόχους σχετικά με το κλίμα και εμείς έχουμε εμπορικές πολιτικές από την άλλη πλευρά, πολιτικές ελευθέρων συναλλαγών, υποβολή ε, τυφλή ε, της εμπορικής πολιτικής στο φιλε, νεοφιλελεύθερο ε, δόγμα ε, και δεν λαμβάνουμε υπόψη τη συμφωνία για το κλίμα. Αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ κακή για τον πλανήτη. Αγνοεί πλήρης την αρχή της προφύλαξης, δεν προβλέπει κανένα περιοριστικό μέτρο, καμία κύρωση σχετικά με την αηφόρο ανάπτυξη και δεν λαμβάνει ουδόλως υπόψη τις κριτικές που εκφέρουμε συνεχώς ε, και εκφέραμε όταν συνάφθηκε η ΣΕΤΑ και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε ένα σημείο που αγνοήθηκε πλήρως το θέμα της αλίας, της αλίας της φάλαινας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ε, ποιο ρόλο ε, παίζει ε, η Ιαπωνία, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα διεθνές μορατόριο και παρόλα αυτά εμείς εξετάζουμε μια εμπορική συμφωνία χωρίς να εξετάζουμε αυτό το θέμα. Για όλα αυτούς τους λόγους η ομάδα μας θα αντιτεθεί σε αυτή την συμφωνία. Αλλά δεν είναι καλή μέθοδος δημοκρατική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει να πει ναι ή όχι μόνον. Και αν έχουμε το θάρρος θα πρέπει να πούμε όχι, διότι σήμερα και με αυτού του είδους της μεθόδου και της, ε, των ευθέρων συναλλαγών ε, που θέτει σε κίνδυνο τις πολιτικές της Ευρώπης ε, θα επιδεινωθεί η κατάσταση και όταν θα το αντιληφθούμε θα είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι εγώ υποστηρίζω στεναρά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Εγώ άλλωστε ε, είμαι και εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη συγκεκριμένη συμφωνία για την ενίσχυση συνεργασίας και θέλω να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που η γρομοδότηση είτε δεν πετυχαίνει σωστά είτε ε, αποσιωπά. Αναφέρεται ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Ωστόσο, Κάθε δισεκατομμύριο εξαγωγών ε, αντιστοιχεί σε 14 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ενισχύει την, την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ. Ρυθμιστική συνεργασία ε, Ένωσης και η Ιαπωνία θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε στενότερα για την ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών ε, και την σύγκληση όταν οι κανόνες μας αποκλίνουν ή είναι πολύ διαφορετικοί. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει η γνωμοδότηση αυτή, ότι ε, δεν υπάρχει πλατφόρμα για την ε, βελτίωση των προδιαγραφών και των προτύπων μεταξύ των δύο οικονομιών των δύο πλευρών. Επίσης, στην γνωμοδότηση δεν αναφέρονται και δεν αιτιολογούνται με στοιχεία επαρκώς διάφορες αναφορές, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός ότι ε, η Ιαπωνία ε, αναφέρεται ότι είναι σημαντικός εισαγωγέα ε, ξυλίας. Δεν είναι. Είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μεγαλύτερο, Υπάρχουν και μεγαλύτερο, όπω είναι η Κίνα, για παράδειγμα. Επίσης, το DPA συνοδεύεται και από SPA, δηλαδή... Ε, προβλέπονται και κοινέ δράσεις για την αντιμετώπιση περιφερειακών αλλά και διεθνών προκλήσεων όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, η αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Οι απόψεις προστατευτισμού που εκφράζονται με αφορμή αυτήν την συμφωνία μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση η οποία θα υποστηρίζει την πρόταση για απόφαση του, του Συμβουλίου για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Ευχαριστώ πολύ και με αυτό ολοκληρώνουμε ε, τον κατάλογο των σκιωδών. Αν θέλει κάποιος άλλος, κάποιο μέλος τη επιτροπή μα να λάβει το λόγο, αν όχι, τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Τσιρούλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Και σας ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις θέλω να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια, ιδίως σε εκείνα ε, που απευθύνθηκαν στην ε, Κομισιόν. Θα ξεκινήσω με το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος που αναφέρθηκε και το ζήτημα της προστασίας των επενδύσεων ως αναπληρωτής επικεφαλής ε, των διαπραγματευτών εγώ συμμετείχα ενεργότατα στις διαπραγματεύσεις και στην εξέλιξή τους και πρέπει να σας πω ότι παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Και το μόνο στοιχείο που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε και αυτό επειδή προσπαθούμε να απαντήσουμε και στον επίγοντα χαρακτήρα που έδωσε ε, το Κοινοβούλιο στο σύστημα ICS, το κάναμε αυτό διότι είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας να διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό, το πώς τα κράτη-μέλη και ε, το Κοινοβούλιο μας ζήτησαν να διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό. Και λόγω αυτής της εντολής δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση αυτή και γι' αυτό και δεν εντάχθηκε σχετικό κεφάλαιο στη συμφωνία. Στόχος μας βεβαίως ήταν να σας παρουσιάσουμε τα όσα είχαμε επιτύχει κατά τις διαπραγματεύσεις στη συμφωνία, αλλά ε, μόλις καταλήξουμε και σε συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων με την Ιαπωνία, βεβαίως αυτή η συμφωνία θα σας δημοσιοποιηθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία βεβαίως. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που γίνεται πάντοτε και με μια πολύ συγκεκριμένη και προβλεπόμενη διαδικασία. Γι' αυτό και υποβάλλουμε τη συμφωνία όσο έχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις, με τις προβλέψεις της συνθήκης, σε εσάς για έγκριση. Και η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει μια, φορά, μια σειρά από πολύ σημαντικά στοιχεία. Ε, η διαφάνεια. Από το πουθενά ήρθε αυτή η συμφωνία ξαφνικά. Όχι. Κάθε άλλο, η συμφωνία αυτή έχει συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και σε άλλες συνεδριάσεις τουλάχιστον 30 φορές στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όλα τα έγγραφα έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, έχει υπάρξει διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών εξασφαλίσαμε το μέγιστο βαθμό διαφάνειας στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις και με αυτό ανταποκριθήκαμε και στο δικό σας αίτημα κατά το περιθόν να εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο διαφάνειας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το κάναμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό Κάναμε διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς, με ενδιαφερόμενους, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με επικεφαλής σε πολλές από αυτές τις συναντήσεις την Επίτροπο Μάλστρομ που ήταν και η επικεφαλής των διαπραγματευτών και στο πλαίσιο των οποίων δόθηκαν σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετείχαν ε, όλα τα στοιχεία που συζητούνταν κατά τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχεδόν μηνιαίως, ίσως κάθε δύο μήνες, σε πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια είχαμε συναντήσεις μαζί σας και πρέπει να σας πω ότι αυτή καθ' αυτή η συμφωνία συμπεριλαμβάνει μια σειρά από στοιχεία που προτάθηκαν από ευρωβουλευτές, από πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Αυτά ως προς τη διαφάνεια. Και επίσης θα έχετε παρατηρήσει ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δημοσιεύονταν εκθέσεις μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων και δημοσιεύονταν και τα κείμενα επί των οποίων είχαν βασιστεί οι συζητήσεις. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει την ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ζήτημα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και του εμπορίου και το αντίστοιχο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναφορές στην ε, τήρηση των ε, περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων, την προστασία των επενδύσεων, την, το σεβασμό στην εργατική νομοθεσία, την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, εταιρική κοινωνική ευθύνη και περιλαμβάνει και μια διαδικασία επίλυσης ε, διαφορών η οποία αποτελείται από διάφορα στάδια, δημιουργία επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βασίζεται και στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια και εντάσσει βεβαίως και ανεξάρτητους φορείς καθώς και διεθνείς φορείς όπως είναι ε, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Και βεβαίως σε όλη αυτή τη διαδικασία εμείς στηρίσαμε την εντολή που λάβαμε καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές που λάβαμε από τα κράτη-μέλη. Και θεωρώ ότι καταφέραμε να διαπραγματευτούμε ένα πολύ ολοκληρωμένο κεφάλαιο στον τομέα αυτό. Όσον αφορά την παράνομη υλοτομία. Σας ευχαριστώ την προσοχή στο γεγονός ότι πρόσφατα η Ιαπωνία ενέκρινε νέα νομοθεσία για την παράνομη υλοτομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τη διαδικασία αυτή. Θα συνεχίσουμε βεβαίω τώρα να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτής της νέας νομοθεσία. Και όχι μόνο προβλέπεται και περιλαμβάνεται συγκεκριμένο άρθρο για την παράνομη υλοτομία που δεν χρησιμοποιεί καθόλου ε, η ποιότερη γλώσσα από ότι αυτή που χρησιμοποιείται σε άλλες συμφωνίες αλλά ταυτόχρονα ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλία εξακολουθεί να ισχύει και με δεδομένη αυτήν την ε, συμφωνία. Θα πρέπει δηλαδή οι εισαγωγέ από Ευρωπαϊκή Ένωση να, να παίρνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν θα εισάγεται παράνομη ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ιαπωνία. Θα συνεχίσουμε μάλιστα και την στενή μας συνεργασία με την Ιαπωνία στον τομέα αυτό για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Άλλα σχόλια. Ιαπωνικά οχήματα. Βεβαίω υπάρχει μια ε, απελευθέρωση στον τομέα αυτών ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οχημάτων και ξέρετε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την τάση που υπάρχει στον κλάδο και στην, στον κλάδο αυτό της οικονομίας. Οδεύουμε προς όλο και πιο καθαρά αυτοκίνητα. Είναι προφανέ λοιπόν ότι πρέπει όλοι μα να είμαστε πιο ανοιχτοί σε καινοτόμα και φιλικά προ το περιβάλλον προϊόντα στο μέλλον. Το γεγονό λοιπόν ότι ανοίγουμε τι αγορέ μα στα Ιαπωνικά αυτοκίνητα θα πρέπει να ε, συνοδεύεται και, να συνεκτιμάται σε αυτό ότι πολλά από αυτά τα ιαπωνικά αυτοκίνητα παράγονται και κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μιλάμε για 2,5 έως 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο. Ακόμη και αν υπάρξει όμως αύξηση των εισαγωγών, καθόλου δεν δίνεται ε, προβάδισμα ή προτεραιότητα σε άλλα αυτοκίνητα πλην των καθαρών αυτοκινήτων στο μέλλον μέσω της συμφωνίας αυτής. Για τη φαλαινοθυρία, βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσιλωμένη και δεσμευμένη στους κανονισμούς και τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των φαλενών. Και βεβαίω υπάρχει αυτό το παγκόσμιο μορατόριουμ το οποίο συνεχίζουμε και ε, στηρίζουμε και εφαρμόζουμε. Συγκεκριμένα στην συμφωνία αυτή η εμπορική φαλαινοθυρία βεβαίως δεν αναφέρεται στην, στην εμπορική μας συμφωνία γιατί ακριβώς δεν, δεν είναι αντικείμενο εμπορίας οι φάλαινε και τα προϊόντα φάλαινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεν χρειάστηκε καθόλου να εντάξουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο στη συμφωνία μας. Παρά την ε, δεδηλωμένη θέληση των Ιαπώνων, πρέπει να σας πω. και βεβαίω καθόλου δεν θα επηρεάσει η σύναψη αυτή τη συμφωνία την γενική μας στάση σε όλα τα διεθνή φόρα όσον αφορά την ε, αντίρρησή μας ε, στη φαλαινοθυρία. Τέλος, ε, αρχή προφύλαξης. Να σας πω για αυτό το θέμα ότι δεν είναι ορθό ότι δεν αναφέρεται καθόλου. Στο άρθρο 16 σημείο 9 αναφέρεται. Και επίσης κατοχυρώνεται η συγκεκριμένη αρχή και στη συνθήκη μας, η οποία βεβαίως και υπερισχύει ως πρωτογενές δίκαιο της συμφωνίας με την Ιαπωνία. Αυτή η αρχή προφύλαξης λοιπόν καθόλου δεν υπονομεύεται ούτε υποσκάπτεται από τη συμφωνία αυτή. Το αντίθετο. Άλλωστε de facto αποτελεί και μία από τις εξαιρέσεις που συνοδεύουν αυτή τη συμφωνία όσον αφορά τους τομείς που δεν καλύπτονται από συγκεκριμένες διατάξεις της συμφωνίας. Φυσικά λοιπόν και η αρχή της προφύλαξης παραμένει στο επίκεντρο και στην καρδιά του δικαιικού μας συστήματος Καθόλου δεν υποσκάπτεται η αρχή αυτή από τη συμφωνία με την Ιαπωνία και βεβαίως εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους και οι κανόνες του ΠΟΕ. οι οποίοι επίσης υπερισχύουν τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Ντροσένσκη δεν ξέρω αν θέλει να πάρει και πάλι το λόγο. Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Θα τα διαβιβάσω όλα αυτά στην κυρία Μελόν. Και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο που μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τις εκθέσεις εξ ονόματο τη κυρίας Μελόν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 5 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΜΒΗ στις 18 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνονται λοιπόν τα σημεία αυτά στην ημερήσια διάταξη και τώρα πάμε στο σημείο 5. Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολή εκθέσεων στον τομέα τη περιβαλλοντική πολιτική. Είναι δικό μου θέμα αυτό. Καταρχάς λοιπόν ε, να πω ότι καλωσορίζω την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευθυγραμμίσει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και να επικαιροποιήσει συγκεκριμένε διατάξεις ε, των οδηγιών που αφορούν ε, τους κανονισμούς και των οδηγιών και των κανονισμών, συγγνώμη, και όπως ξέρετε οι προτάσεις αυτές απορρέουν από ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα δράσης για την ευθυγράμμιση των εκθέσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ένα από τα αποτελέσματα του ελέγχου που έγινε βάσει του fitness check για την πολιτική αυτή και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώνει την πρόσφατη απόφαση για τους διαδικαστικούς κανόνες για τις ε, εκθέσεις σε περιβαλλοντικά θέματα. Εγώ υποστηρίζω βεβαίω το στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια, να βελτιώσουμε την συλλογή στοιχείων για τι μελλοντικέ αξιολογήσει και να απλοποιήσουμε και το διοικητικό άχθο και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, υπέβαλα κάποιε τροπολογίε με στόχο να βελτιώσουμε την νομοθετική πρόταση που θα πρέπει να εξυγχρονίσει την διαχείριση των ε, πληροφοριών και να μειώσει το διοικητικό άχθο. Η πρόταση που έγινε να υπάρχει πιο διάφανη πρόσβαση σε σαφείς περιβαλλοντικές πληροφορίες για αρκετούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένου και του κοινού, που συμβάλλει μεταξύ άλλων και στο στόχο προτεραιότητας 4. Για παράδειγμα, ε, αρκετές ε, τροπολογίες αφορούν τους ορισμούς ε, αρκετών όρων σε βασικές πράξεις και δίνουν και κάποιες λεπτομέρειες για κάποιους όρους και στόχο έχουμε να έχουμε καλύτερη συνοχή και απλούστευση του κειμένου και ελπίζω να διευκρινίσουν περισσότερο τα πράγματα. Επίσης, προσπάθησα να βελτιώσω το ρόλο του συνομοθέτη και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και να διευκρινίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την όλη διαδικασία υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης. Όσον αφορά την οδηγία 35, για την περιβαλλοντική ευθύνη που αφορά την πρόληψη και τις περιβαλλοντικές ζημίες. Πιστεύω ότι τα αναλυτικά κριτήρια είναι απαραίτητα σε αυτή την περίπτωση να ε, έχουμε ταξινόμηση της ε, κλίμακας της περιβαλλοντικής ε, ζημίας και στην περίπτωση της οδηγίας 63 για την προστασία της χρήσης ζώων για επιστημονικούς λόγους ε, προτείνω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να δημοσιεύει, αλλά να ενημερώνει τακτικά για την ε, συνολική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη για την, ε, τον κανονισμό 166 για τους ε, ρηπογόνους παράγοντες ε, και το σχετικό μητρό. Προτείνω μια σαφή προθεσμία υποβολής εκπαίδευσης από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δίνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό. Για τον 995 για τα προϊόντα ξυλία και την ξυλία ε, και τη διάθεσή του στην αγορά, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τις νομοθετικές προτάσεις που γίνονται σε κάθε νομοθετική θητεία και να μειώσει και την ε, περίοδο αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα 6 στα 5 χρόνια. Τέλος, έχω προτείνει κάποιες αλλαγές όσον αφορά κάποιες διατάξεις που αφορούν ε, τη χρήση της ε, ρυθμιστικής διαδικασίας για τον έλεγχο στις βασικές πράξεις. Κατά την άποψή μου, οι διάφορες διατάξεις που προτείνονται εδώ θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την συνθήκη της Λισαβόνας και εδώ ζητώ να χρησιμοποιούνται πράξεις κατεξουσιοδότηση σε κάποια άρθρα συγκεκριμένων πράξεων ε, που αναφέρονται στην πρόταση. Ελπίζω αυτό να διευκρινίσει περισσότερο ε, τις εξουσίες που εκχωρούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δύο συνομοθέτες. Τώρα, όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβένας και την χρήση πράξεων κατεξουσιοδότησης, ε, όχι μόνο θα επικαιροποιήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα βελτιώσει την όλη διαδικασία υποβολής εκθέσεων και εποπτείας. Αυτά λοιπόν εν είδη σύντομη παρουσίαση για κάτι το οποίο είναι αρκετά τεχνικού χαρακτήρα και νομοθετικού. Ε, Βασίζομαι βεβαίω στην υποστήριξή σα για περαιτέρω βελτίωσή του. Να στραφώ λοιπόν στους κοιόδης ε, εισηγητέ. Ο κύριος Παολούτσι καταρχάς. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου Ευχαριστώ πολύ γιατί όσα κάνατε. Πρόκειται για μια πολύ αναλυτική δουλειά. Εμείς από πλευράς μας επαληθεύουμε ότι η διάθεση των ε, στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη-μέλη και η δημοσίευσή τους ε, πρέπει να εξασφαλίζεται στις διάφορες νομοθετικές πράξεις και ή δυνατόν για αυτό το συγκεκριμένο σημείο θα κάνουμε και πιθανές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Mr. Pieka. Uh, no. Oh. Mr. Martinez. Ο κύριος Μαρτίνεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι που η πρώτη συνεδρίαση μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι εδώ στην Επιτροπή σας, την οποία απολαμβάνω πάντα. Επειδή η έκθεση αυτή είναι δική σας, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω λοιπόν για ό,τι έχετε κάνει. Ε, και τα εκτιμούμε ιδιαίτερως. Θα γνωρίζετε βεβαίως ότι η ομάδα μας ε, είναι πάντα υπέρ της μείωσης ε, των κανονισμών για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις, επομένως πρόληψη περισσότερων εργαζομένων και να βελτιώσουμε και την οικονομία. Και ε, επίσης τα περισσότερα χρήματα τα οποία δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα θεσμικά όργανα για τη συλλογή δεδομένων, σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα δώσουν για άλλους σκοπούς. Θα πρέπει λοιπόν πάντα να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πιέσεις προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κατά πόσον, ε, κατά πόσον θα μπορούσαμε να δαπανούμε αυτό το χρόνο αλλιώ. Έχω βέβαια κάποια πράγματα και θα ήθελα να τα επισημάνω και να πω ότι μας ανησυχούν. Πρώτον, δεν καταλαβαίνουμε λίγο τη λογική. Γιατί ε, υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις για την Οδηγία 2004-35 και τον Κανονισμό 166-2006. Μπορεί να θεωρείται απαραίτητο, αλλά θα θέλαμε κάποιε διευκρινήσει για ποιο λόγο θεωρείται απαραίτητα πριν μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε. Και δεύτερον, παρά το γεγονό ότι εκτιμώ ιδιαίτερο στα σχόλιά σα για την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τα πάντα ευθυγραμμίζονται με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε βάσει ποια λογική ε, το άρθρο 18α, η πράξη κατεξουσιοδότηση, περιλαμβάνονται εδώ. Θα μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε μεν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρω ε, βάσει ποια λογική γίνονται όλα αυτά και θα θέλαμε κάποιε περαιτέρω εξηγήσει πριν αποφασίσουμε. Συνολικά υποστηρίζουμε την έκθεση, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και ε, υποστηρίζουμε και τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή η απλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βύση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ε, αρχίζουμε σήμερα το απόγευμα. Ε, μιλώ εκ μέρους Φρεντερικ Φρεντερλέ που είναι σκιώδης ε, Επίσης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για να μειωθούν οι δαπάνες για τους ενδιαφερόμενους και για να υπάρχει ε, αποτελεσματικότερος τρόπος συλλογής χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά ε, μέσα για τα δεδομένα μεταξύ των τροπολογιών που υποβάλλατε κυρία υποστηρίζει ε, το να υπάρχει πρόσβαση πιο διαφανής για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες για τους ενδιαφερομένους και την πρόθεση να υπάρξει καλύτερη ε, συνέπεια ε, και να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια στην πρώτη μεταβολέσα ε, που πρότεινε η εισηγήτρια για να ενισχυθεί ο ρόλος του συνομοθέτη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διευκρινιστεί ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην υποβολή εκθέσεων και στην παρακολούθηση για την ομάδα μας στην ΑΛΔΕ νομίζω ότι είναι σημαντικές οι εκθέσεις για την νομοθεσία βλέπουμε πώς εφαρμόζονται η νομοθεσία και αν πληρεί τους στόχους και δίνει πληροφορίες για τους πολίτες παραμπτώς χάρη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας κλπ. Επίσης μειώνει τον φόρτο το διοικητικό για τα κράτη-μέλη, αυξάνει την διαφάνεια και εξασφαλίζει ότι θα έχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται το ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον στόχο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Φρεντερικ, σας ευχαριστεί για την, ε, την εργασία σας και χαίρετε για την συνεργασία μαζί σας, κυρία Κολέτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε βέβαια το βασικό είναι να ξέρουμε ποια είναι η ποιότητα του αέρα, η ποιότητα του ύδατος που πίνουμε, των λιμνών κλπ. Θέλουμε ενημερωμένες πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος και αυτός είναι ο βασικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Αλλά έχουμε και τον ρόλο της Κομισιόν που να επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Χαιρετίζουμε την εκθεσή σας και θα τονίσω, με υπογραμμίσω ε, μερικές συνεισφορές που βρίσκουμε ότι προτείνεται για τεχνικές ε, τροποποίησεις ε, στην Κομισιό που αναφέρατε στην παρέμβασή σας τον, θέλετε να ενισχύσετε τον ρόλο του Οργανισμού Περιβάλλοντος ε, σε όλο το θέμα της υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης ευθυγραμμίζοντας ε, τις υποχρεώσεις ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει, να αναθεωρεί ή να τροποποιεί τα διάφορα σημεία. Επίσης χαίρομαι ε, για τις διάφορες τροπολογίες και σας ευχαριστώ για την εργασία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο για το θέμα αυτό. Mr. Eck, you indicated you want to speak. Κύριε Εκ, ζητήσατε το λόγο. Please. Danke, Frau Präsidentin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς μόλις ήρθα, δεν ξέρω ποιο θέμα συζητούμε. Συγγνώμη, ναι. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία. Uh, συζητούμε το θέμα 5, κυρία Εκ. Και είστε σκιώδης. Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σημείο 7 ρωτάει ο κύριος Εκ. Όχι 5 απαντάει η πρόεδρος. Όχι, γι' αυτό το θέμα δεν ήθελα να πω κάτι. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Εκ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να αναλάβετε τη σύνταξη έκθεσης για αυτό το πολύ περίπλοκο νομοθέτημα. Ακούσαμε με προσοχή την περιγραφή του εισηγητή σας και τις παρεμβάσεις των σκιωδών. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή σας κάποιες γενικές αρχές που ενέπνευσαν την Κομισιόν κατά τη σύνταξη της πρότασης αυτής. Και θεωρούμε ότι κάποιες από τις αρχές αυτές και κάποιοι από τους στόχους αυτούς απαντούν και σε ορισμένες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ένας βασικός στόχος μας ήταν να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν τους πολίτες μας, όχι μόνο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι πολύ σημαντικό οι περιβαλλοντικές πληροφορίες, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση του περιβάλλοντος, να είναι γνωστές και στους πολίτες και να μην κατευθύνονται μόνο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ε, άλλα πολιτικά όργανα. Αυτό ε, θα ενισχύσει την επικουρικότητα και τη λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να εξάγει και συμπεράσματα με βάση τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών. Δεύτερη γενική αρχή που μας ενέπνευσε στο έργο μας ήταν η ανάγκη να βασίζεται η χάραξη πολιτικής σε στέρεα στοιχεία. Και έτσι, όπως είπε και ένας από τους σκιώδεις εισηγητές, Θέλω να σας διαβεβαιώσω και τον ίδιο και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας ότι παρά το γεγονός ότι η πρότασή μας επιχειρεί να ελαφρύνει το διοικητικό φόρτο είμαστε άτεγκτοι στην προσπάθειά μας να μην αφαιρέσουμε από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πληροφορίες που σχετίζονται με το πώς υλοποιούνται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών επιτόπου. Μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης ήταν επίσης ένας από τους σημαντικότερους στόχους που είχαμε κατά νου, κατά τη σύνταξη της πρότασής μας. Η χρήση λοιπόν των νέων τεχνολογιών συμβαδίζει με τη μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας ήταν όρημη η απέτηση αυτή και όπως έχουμε κάνει και με άλλες ευκαιρίες, ευκαιρίες στην ε, περιβαλλοντική πολιτική προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τους δορυφόρους, τις τεχνολογίες προφορικές προκειμένου να βοηθήσουμε τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να μπορεί να σχηματίσει μια συνολικότερη εικόνα για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Και αυτό διότι πολλές φορές πνιγόμαστε στις λεπτομέρειες διαφόρων διοικητικών ρυθμίσεων και διατάξεων και δεδομένων και ταυτόχρονα χάνουμε τη γενική εποπτεία, τη γενική εικόνα που δεν πρέπει κανείς να χάνει ποτέ από την προσοχή του. Γι' αυτό και θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή σας να προχωρήσει στο έργο της, όπως έχετε ήδη βεβαίως κάνει κυρία Πρόεδρε και όπως ήδη αναφέρετε στην ε, έκθεσή σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι έχετε ενημερώσει, επικαιροποιήσει τον συσχετισμό μεταξύ των διατάξεων της πρότασης που υπέβαλε η Κομισιόν. Ένα ε, σχόλιο φορούσε τη σχέση τη συγκεκριμένη πρόταση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόταση που έχουμε υποβάλει συνάδει απολύτως με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η δική σας έκθεση ακριβώς ενισχύει αυτόν τον συσχετισμό. Η ετήσια έκθεση που υπέβαλε η Κομισιόν πριν από κάποια χρόνια αφορούσε την ευθυγράμμιση του ευρωπαϊκού δικαίου με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και δεν έχει εγκριθεί πλήρως από τους συνομοθέτες. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό και παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εμείς υποβάλλουμε αυτήν την νομοθετική πρόταση και αυτές τις λύσεις που θεωρούμε ότι ευθυγραμμίζονται με τις βασικές αρχές της πρότασης Omnibus για τη λισαβονοποίηση. Και στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε να προσέχουμε και να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρχει απόκληση μεταξύ αυτής της πρότασης και της πρότασης Omnibus για την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και ένα τελευταίο σχόλιο να κάνω κύρια Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, πρόσθετες τροπολογίες που έχετε εντάξει στην έκθεσή σας όσον αφορά την, οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης που απαντούν στον έλεγχο καταλληλότητας που ε, διεξήγαγε η Κομισιόν πριν από 2-3 χρόνια όσον αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία και ο οποίος έλεγχος έδειξε ότι το μέσο αυτό προκειμένου να μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χρειάζεται περισσότερες προφορίες περισσότερα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη για κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται στα κράτη-μέλη και σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Και με αυτό απαντώ και σε μια άλλη παρατήρηση που έγινε από σκιώδη εισηγητή να σας πω ότι δεν προσθέτουμε πουθενά διοικητική επιβάρυνση. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις επιπλέον που προκύπτουν από την οδηγία ε, για την περιβαλλοντική ευθύνη και εμείς στην ουσία ε, ερχόμαστε και απαντούμε στην αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή και την εκτέλεση αυτής της οδηγίας. Αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν ε, μας αποδεικνύουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να χαράξουμε αποτελεσματικότερες πολιτικές. Και γι' αυτόν τον λόγο ε, επιμένουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, υπάρχουν αυτές οι πρόσθετες διατάξεις ακριβώς γιατί θα μας αποφέρουν πολύ σημαντικά και θετικότατα αποτελέσματα. Γι' αυτό και θα ήθελα να καλέσω και τη δική σας Επιτροπή να υποστηρίξει αυτήν την τροπολογία. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος για το ενδιαφέρον που έχετε εκφράσει στο θέμα αυτό και για την υποστήριξή σας και νομίζω ότι με τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας θα καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Θα απαντηθούν οι ανησυχίες και τα ερωτήματα που εκφράστηκαν. Ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 4 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. 10 και 11 Οκτωβρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Ένβη και με αυτό ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό και περνάμε στο σημείο 6. Μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Φάκελος συναπόφασης θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης που έχει συντάξει η κυρία Ρης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα βεβαίως ε, σήμερα μπαίνουμε στην ουσία του θέματος, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαντς, όταν ήρθε τον Ιούνιο να συνομιλήσει μαζί μας, ε, νομίζω ότι ε, το θέμα είναι επίγον. Νομίζω και όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την σημασία να κλείσουμε το θέμα πριν από τις εκλογές. Μια πρόταση οδηγίας και μια συζήτηση σήμερα που βεβαίως ε, δεν, δεν δικάζουμε τα πλαστικά. Τα πλαστικά τη δεκαετία του 50 ήταν επανάσταση ε, που έφεραν αλλαγές στα πάντα, στις πρακτικές, στις αντικείμενα και στις συμπεριφορές. Εναπόκειται σε άλλους ε, να ασχοληθούν με το θέμα, αλλά εμείς οι νομοθέτες πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση, έναν απολογισμό διότι πάρα πολλοί πεθαίνουν από αυτό. Έχουμε μερικούς αριθμούς που δεν αμφισβητούνται, δεν πρόκειται να τους επαναλάβω εδώ. Αυτό που μας απασχολεί τώρα αναφέρεται στα πλαστικά μιας χρήσης, ε, δηλαδή τα ε, καλαμάκια, οι αναδευτήρες, ε, τα, τα κυπελάκια, τα μαχαίρια, τα πυρούνια, όσα χρησιμοποιούμε μία λεπτό, δύο λεπτά και μετά τα πετάμε ένα λεπτό μετά. Βεβαίως 86% των πλαστικών απορριμμάτων που βρίσκουμε στις παραλίες στην Ευρώπη είναι ακριβώς αυτά τα αντικείμενα μιας χρήσης ε, και από τα 26 εκατομμύρια ε, τόνους απορριμμάτων από τους Ευρωπαίους μόνο ένα μικρό μέρος, 4% ε, είναι ανακυκλώσιμα πλαστικά. Δεν μπορεί να διονυστεί αυτή η κατάσταση άκουσα μερικούς ε, που λένε ότι πρέπει να ε, εξετάσουμε περισσότερο το θέμα, αλλά ε, έχουμε την απόρριψη στη θάλασσα πολλών από αυτά τα πλαστικά απορρίμματα και η Ευρώπη δεν έχει leadership ως προς το ε, θέμα αυτό. Στο Ρίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για, την, ε, για τον αγώνα κατά ε, της αναθέρμανσης του κλίματος και σήμερα πρέπει να κάνουμε το ίδιο για τα πλαστικά απορρίμματα. Εμεί, εγώ συμμερίζουμε τις μεγάλες γραμμές της πρότασης της Κομισιόν για τα μακροπλαστικά ε, και επίσης το υλικό αλληλείας που είναι υπεύθυνο για μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων και ευχαριστώ τους ε, ε, αντιπροέδρους Τίμερσαν Κατάινεν και τον Επίτροπο τον Αρμόδιο θα πρέπει να απαγορεύσουμε εκεί όπου είναι δυνατόν τα καλαμάκια και άλλα διότι έχουμε εναλλακτικέ λύσεις από μπαμπού, από καλάμια και που δεν κοστίζουν ακριβά αυτά τα καλαμάκια και για τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουμε μια δέσμη μέτρων ο λιγότερο ε, ρίζοσπαστική με ένα στόχο ε, μη ποσοτικοποιημένο για τα βεβαίως τους περιέκτες τροφίμων για τα κυπελάκια που έχουμε στο άρθρο 4 μια υποχρέωση σήμανσης ε, για ε, τις διάφορες τα μαντιλάκια, τα υγρά για τις σερβιέτες υγιεινής και να ευαισθητοποιήσουμε τους παραγωγούς. Στην αξιολόγηση αντικτύπου σελίδα 46 ε, βλέπουμε το κόστος οφέλος ανάλογα ε, με διάφορες επιλογές, ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας που θα πρέπει να προσδιορίσουμε και ζητώ από την ε, Κομισιό να τα λάβει αυτά υπόψη Ακούω τις κριτικές για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δημοσιοποιήσουμε ε, την μελέτη των συμβούλων, την μελέτη αντικτύπου. Επανέρχομαι στο σενάριο αυτό, στο σενάριο Γ, το οποίο αντιστοιχεί στην επιλογή την πολιτική που έκανα στην εισήγηση αυτή για να αποφύγουμε ζημίες περιβαλλοντικές, των οποίων το κόστος θα είναι 22 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030 και θα μπορούν 6 δισεκατομμύρια να εξοικονομηθούν. Κόστος για τους παραγωγούς 3,2 δισεκατομμύρια ε, και η τιμή θα είναι πολύ ψηλότερη για την βιομηχανία ε, την ευρωπαϊκή. Ε, σχετικά με τα πλαστικά τα οποία απορρίπτονται. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πέρασαν από τη μία μέρα στην άλλη ε, στην ιστορία μας σε μια άλλη συμπεριφορά ε, και απέριψαν τις ελαφρές πλαστικές σακούλες και μπορούμε λοιπόν να έχουμε άλλες επιλογές, άλλες συμπεριφορές. Βεβαίως διαρωτώμε για την επέκταση του συστήματος της υπευθυνότητας των παραγωγών έτσι όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 1 και 2. Είναι θα πρέπει οι παραγωγοί να πληρώνουν ε, για τον καθαρισμό των ποταμών, αυτοί που παράγουν τα υγρά μαντιλάκια και τις σερβιέτες. Θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί. Υπάρχει συνέπεια νομική ε, και έχουμε την τροπολογία 31 που υπενθυμίζει ε, στα πλαίσια της οδηγίας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεχθεί μέχρι την διευρυμένη ευθύνη παραγωγού μέχρι τις 31 ε, για αυτήν την τροπολογία όπως και για το σύνολο των τροπολογιών της εισήγησής μου εργάστηκα με τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο άρθρο 4 για την μείωση κατανάλωσης ε, των περιεκτών τροφίμων και των πλαστικών κυπέλων μου φαίνεται ότι η διατύπωση είναι πάρα πολύ ασαφής, επιδέχεται πολλές ερμηνείες χωρίς μεθοδολογία και χωρίς να έχουμε πολιτικές ποσοτικοποιημένες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό στον τροπολογία 23 υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και μια διαδικασία. Θα έχουν τέσσερα χρόνια για να έρχουν σχέδια εθνικά μείωση με τον έλεγχο της Κομισιόν. Όσον αφορά τις φιάλες τώρα, ε, τις ε, φιάλες, ε, τα καπάκια, τα καλύματα, είναι η πρώτη κατηγορία που βρίσκουμε στην θάλασσα. Εν πέμπτον είναι οι φιάλες. Τροπολογία 27, ένα στόχο να μειώσουμε κατά 25% για το 2025. Είναι μια δέσμευση του τομέα και υπάρχει ήδη leaders, πρωταθλητές στον τομέα που αναφέρουν 100% ανακύκλωση για αυτή την ημερομηνία. Επίσης, περιέλαβα ένα στόχο ανακύκλωσης για τα υλικά αλίας για το 2025, είναι η τροπολογία 33 και εδώ ο στόχος, ο ποσοτικός είναι ρεαλιστικός. Η Ισλανδία έχει 85% ε, που ανακτώνται από τα δίκτυα και τα υλικά αλίας. Για δύο άλλα θέματα έχω στόχο υψηλότερο από το Κομισιό ε, τα φίλτρα τα πλαστικά τσιγάρων ε, που δεν καλύπτονται από την οδηγία, ε, από την κυρία Όγκεν. 500 και 1000 λίτρα ύδατος ρηπαίνονται και έχουμε μια μελέτη του 2014. Βλέπουμε λοιπόν τις επιπτώσεις αρνητικέ πάνω στην υγεία και πάνω στο περιβάλλον. Και εδώ τα θέματα αυτά, η κυρία Γκροστέτ και άλλοι συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Με την οδηγία 2013 για τον καπνό ε, ε, καταθέτω λοιπόν την τροπολογία 25 και εκτός από την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης ε, για τους παραγωγούς καπνού και σιγαρέτων θα πρέπει να μειωθεί η χρήση των φίλτρων των πλαστικών 80% μέχρι το 2030. Και εδώ εργάστηκα με εμπειρογνώμονες από το τμήμα ε, ελέγχου του καπνού ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Έχουμε εναλλακτικές ε, λύσεις και είχαμε μια αναβολή για τους παραγωγούς. Θα πρέπει λοιπόν να απαγορεύσουμε τα υλικά αυτά που δεν ε, ε, περιελαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας. Θα πρέπει να υπάρχει μία εξαίρεση ε, για λόγους υγιεινής. Βλέπω ότι έχω περίπου εξαντλήσει τον χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Περιμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις και τις βελτιώσεις που θα προτείνουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κυρία ε, Ο λόγος του ο Καρλ Χάινς Φλόρενς καταρχάς. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρίς, σας συγχαίρω για το γεγονός ότι υπό αυτή την πίεση της κοινή γνώμης αλλά και σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταφέρατε να συντάξετε αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι ε, είναι χαρακτηριστικό της ποιότητας που έχετε ως πολιτικού. Θέλω να ε, να μην επαναλάβω πολλά από αυτά που είπατε, αλλά όποιος δεν έχει καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω όσον αφορά τα σκουπίδια στις θάλασσες, θα ήθελα να τον παροτρύνω να εγκαταλείψει την πολιτική πραγματικά. Δεν είναι δυνατόν να πάρει άλλη αναβολή ή να πάρουν άλλη αναβολή οι προθεσμίες που έχουμε θέσει. Και αυτό δεν αφορά μόνο με μονομένα προϊόντα όπως ε, τα προϊόντα μίας χρήσης, πακέτο, καφέ, φαγητό, στίκ που καθαρίζετε τα αυτιά σας. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική μεταστροφή. Και αυτό αφορά και τις γόπες των τσιγάρων. Αν σκεφτείτε πόσα χρήματα δαπανώνται για να, καθαρίζεται, να καθαρίζονται δισεκατομμύρια λίτρα νερού που έχουν δηλητηριαστεί από γόπες τσιγάρων που βρίσκονται παντού, στους δρόμους μας, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Γιατί, γιατί κακομαθημένοι πολίτες δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα τασάκια που τους προσφέρονται. Είναι ανάγωγοι άνθρωποι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι της ηλικία μου, δεν μιλάω μόνο για την νεολαία. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας στα περισσότερα από αυτά που είπατε. Δεν πρέπει όμως κάποια στιγμή να γίνει μια έκκληση προς τους πολίτες να μαζεύουν τα σκουπίδια τους από τα πάρκα. Είναι δυνατόν να παίρνει ο άλλος σοκολάτα Μάρς και να πετάει το χαρτάκι κάτω και μετά να μετακυλίεται το κόστος αυτό στους πολίτες μας γιατί πρέπει να προσλαμβάνουμε εταιρείε καθαρισμού των πάρκων. Ειλικρινά πείτε μου, οδεύουμε στη σωστή κατεύθυνση. Εμένα γενικά οι απαγορεύσει δεν μ' αρέσουν. Όμως πρέπει να εκπαιδεύσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες μας. Πραγματικά, άμα δείτε τους δρόμους των πόλεών μας, κάθε Κυριακή πρωί, ε, δεν μπορούμε να, να καθιστούμε υπεύθυνε τώρα τις καπνοβιομηχανίες για την κατάσταση που επικρατεί. Η κοινωνία φταίει. Αυτά που είπατε για το χαρτί υγείας είναι σωστό, αλλά υπάρχει, και χαρτί υγείας το οποίο δεν περιλαμβάνει ε, συνθετικές ουσίες. Πώς ακριβώς θα γίνει η ε, διάκριση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συζήτηση καλώς ξεκίνησε, γιατί από αυτή τη συζήτηση θα προκύψουν μαζικής κλίμακας καινοτομία. Πιστέψτε με, καλαμάκια και ε, βοηθήματα ε, για να καθαρίζει κανείς τα αυτιά του θα εξαφανιστούν σε λίγα χρόνια. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχω τρία εγγόνια. Τι θέλετε τώρα να τους πω, ότι δεν μπορούν να πετάξουν το χαρταϊτό τους που είναι παραδοσιακό έθιμο στη Γερμανία ή τέλος πάντων ένα μπαλόνι, δεν μπορώ να τους αγοράσω λόγω του ότι είναι πλαστικό. Ε, δεν γίνεται, εντάξει. Αυτό που μπορώ να τους πω είναι να μην, να μην σκάσει τον μπαλόνι και να αφήσουν το σκουπίδι κάτω. Ναι, φυσικά, να πούμε στους γονείς, άμα σκάσει τον μπαλόνι, να το πετάξουν στο τενεκέ και όχι στο δρόμο ή στο πάρκο. Όμω, φοβάμαι πολύ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με σοβαρότητα προβλήματα. Η Ευρώπη μπορεί και να διαλυθεί με όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και εμεί τώρα καθόμαστε και ασχολούμαστε με την επισήμανση των παλωνιών. Τι να σα πω, ευχαριστώ. Κύριο Περούτσι. κύριο Παολούτσι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ, όπω και ο προλαλή σα συνάδελφο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρή ε, για την εξαιρετική τη δουλειά. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να ενισχύσουμε τα μέτρα τα οποία αφορούν ε, τις, πλαστικές, ε, τις ελαφριές πλαστικές αξικούλες και τις γόπες από τα τσιγάρα και πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και τα μέτρα τα οποία αφορούν ε, τα διάφορα πακέτα γλυκά και πατατάκια και ε, τις συσκευασίες, πλασ, πλαστικές συσκευασίες για παγωτά. Πιστεύω ότι όπως είναι γραμμένη η οδηγία δεν είναι παρκώς ε, ακριβής και θα πρέπει να τη βελτιώσουμε με ελάχιστους κανόνες, ε, ε, διάφανους τρόπους υπολογισμού και πιο καλά χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά την ευθύνη των παραγωγών, πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε όπως κινηθήκαμε αυτούς τους μήνες και με τα όσα έγιναν για την κυκλική οικονομία. Δηλαδή θα πρέπει να προβλέψουμε συμβολή η οποία θα είναι ανάλογη με το προϊόν. Όσο πιο εύκολα μπορεί κάποιος να ανακυκλώσει και να επισκευάσει ένα προϊόν, λιγότερα πρέπει να συνεισφέρει ο παραγωγός και όσο περισσότερο είναι, είναι μεγαλύτερη συμβολή ε, του παραγωγού. Όσον αφορά την αλληλεία, πρέπει να κινηθούμε για να έχουμε μία συμμαχία με τους αλληλείς, για να είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στην όλη αυτή διαδικασία. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ε, τεράστιες διαπάνες για παθητική ε, ε, αλληλεία που γίνεται από τους αλληλείς και θα πρέπει για κάποια αλληλευτικά προϊόντα να έχουμε κάποιες ε, δυνατότητες προφύλαξης, ε, αποζημίωσης ε, κλπ. Και γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και να προτείνουμε μέτρα ενίσχυσης της οδηγίας όσον αφορά την προσπατασία των θαλασσών και των ακτών, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην περιπλέξουμε και χωρίς λόγο τη ζωή των πολιτών. Για παράδειγμα, Κάποια χρήσης ε, πλαστικά μια χρήση ε, στα νοσοκομεία, σε λέσχες, σε κλειστά κυκλώματα, εκεί θα πρέπει να το σκεφτούμε ίσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κάποιο ότι αυτά τα ε, προϊόντα μιας χρήσης δεν μπορούν να είναι από βιοδιασπόμενο πλαστικό. Πιστεύω όμως ότι η δουλειά που γίνεται είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριο Ντέμεσ Μάκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυκλική οικονομία είναι το νήμα της στάθμης που διέπει όλες τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ε θα αποτελέσει και το βασικό ε, θέμα συζήτησης στη στρατηγική για τα πλαστικά στην Ολομέλεια. Εγώ προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα και πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της νομοθετικής διαδικασίας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι είδατε την εξαιρετική ε, ταινία στο facebook έχει γίνει και viral και λέγεται «Η βίβλος των ζώων» και αφορά μια παραλία, νομίζω στην Ινδία, η οποία είναι απόλυτα καλυμμένη από πλαστικά, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Και ε, Κάποιο δεν αντέχει, προσπαθεί να τα καθαρίσει και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τα κάνει από μόνος του, καλεί τους φίλους τους και τελικά όλη η τοπική κοινότητα συμμετέχει σε αυτό τον καθαρισμό της παραλίας. 400.000 ε, ε, ε, χιλιάδες περίπου τόνοι πλαστικών και μετά από μερικές μέρες ως εκθαύματος αρχίζει να φαίνεται η αμμουδιά στην παραλία και αρχίζουν να έρχονται και πάλι χελώνες για να γεννήσουν τα, τα αυγά του στην παραλία. Είναι ένα φανταστικό όραμα της μάχης κατά των πλαστικών. Βέβαια θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι έγινε αργότερα, τι έγινε με αυτούς τους 4.200 τόνους πλαστικού που συνελέγησαν εκεί. Ε, όπως γνωρίζουμε βεβαίως, ε, τα περισσότερα τα σκουπίδια ε, πετιώνται στην Ινδία, δεν υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης ε, και πολλά από τα πλαστικά ουσιαστικά χωματερή ξαναβρίσκονται στη θάλασσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίλυσή του. Το να καθαρίζουμε απλώ όμω τα απόβλητα δεν αποτελεί λύση. Θα πρέπει να σκεφτούμε από πού προέρχονται από αυτά τα απόβλητα και κυρίω να υπάρχει μια προσέγγιση για την όλη παραγωγή και αλυσίδα κατανάλωση για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το μέγεθος ε, της παραγωγής αυτών των πλαστικών. Και με αυτό έρχομαι και στην πρόταση τη Οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή γι' αυτό και την κυρία Ρή, την εισηγήτρια, να την ευχαριστήσω κιόλα για την επικοδομητική και ταχύτατη προσέγγιση της. Πιστεύω ότι μπορούμε σύντομα να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Ε, είχαμε και καλές καλοκαιρινές διακοπές και μπήκαμε κατευθείαν στη δουλειά. Καταρχάς θα ήθελα να πω τα εξή. Από ό,τι κατάλαβα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, επικεντρωθεί στα πρώτα δέκα πιο κοινά πλαστικά, διότι κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να είναι λίγο πιο σαφής ο στόχος της οδηγίας. Επίσης, ε, τι γίνεται με το θέμα για τα πλαστικά μια χρήση. Ε, ε, πρότεινε κάτι η συγγήτρια, θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια πρόταση μέσω τροπολογία. Την περασμένη Παρασκευή επισκέφθηκα ένα μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών εδώ στη Φλάνδρα και γνώριζαν πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν για την ε, μείωση των αποβλήτων από πλαστικά. Και επίση υπάρχει και η αρχή του ρηπαίνων πληρώνω, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και εδώ τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται με διάφανο τρόπο και να είναι και αποτελεσματικά ως προς το κόστος των όσων δαπανώνται. Και εκεί που ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα είναι ε, το μάρκετινγκ, η διάθεση στο εμπόριο. Ε, υπάρχει μια... Ε, ε έκκληση για να χρησιμοποιούμε εμπορικά σήματα για βιώσιμες συσκευασίε, ε, βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης. Νομίζω αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε στο άρθρο 10. Τέλος, εμείς ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι δημόσιες αρχές ε, και οι κυβερνήσει, θα πρέπει να δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Ε, για τον ορισμό στο άρθρο 4 θα ήθελα να ρωτήσω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρεστε σε ουσιαστική προστασία γιατί δεν ε, ε, έχει δώσει στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Η κυρία Αρής πρόσθεσε κάποια νέα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι άποψη έχουν αυτοί για αυτές τις προτάσεις. Μετά, οι απαιτήσει του άρθρου 7. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί να επιτευθεί το άρθρο 7 βάσει των όσων προτείνονται. Και επίσης, ε, χαρτόκουτα για την ε, πλαστική επικάλυψη. Αυτά θα θεωρούνται ως πλαστικά μιας χρήσης. Μπορείτε να με το εξασφαλίσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ακούσω και τι άλλο έχουν να πούν οι συνάδελφοι και να εργαστούμε επικοδομητικά για την επίλυση. Ευχαριστώ η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι όταν εγώ υπέβαλα την πρόταση για τις πλαστικές σακούλες πριν από πέντε χρόνια, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, ε, μάλλον υπεροψία θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Ο κύριος Τίμπερμανς είπε ότι η πρόταση θα ήταν τόσο περίπλοκη στην έγκρισή της, ιδιαίτερα με τον τρόπο με τον οποίο από τους πρασίνους, που θα ήταν σχεδόν αντίνο αδύνατον. Άκουσα πολλά τότε πριν από πέντε χρόνια και με αυτό στο νου μου, μου φαίνεται εξαιρετικό ότι αυτή τη στιγμή πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε μια εξαιρετική πρόταση και ο κύριος Τίμερμαντς είναι ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς που μετανόησε και θα τον δεχτούν με ανοιχτές αγκάλες στον παράδεισο. Είναι εξαιρετικό το ότι έχουμε αυτή την τόσο καλή πρόταση για τα πλαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι θαυμάσιο να αλλάζει κάποιο γνώμη και να βρίσκει το φως του. Και ξέρω ότι στη χώρα του Τίμερμαντς, ε, στις κάτω χώρες, η πρόταση για τα πλαστικά ήταν ε, μεγάλη επιτυχία. Τώρα, προς την κυρία Ρης, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την τεράστια προσπάθεια που κάνετε. Όλοι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να προχωρήσει η πρόταση αυτή, διότι έχουμε μπροστά μας και εκλογέ. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή συγκυρία για μας, ε, για να γνωρίζουμε και σε τι εστιάζουν οι πολίτες. Και μεταξύ μας, η πολιτική για το κλίμα μπορεί να μην είναι ε, η πρώτη απόλυτη προτεραιότητα, αλλά σίγουρα τα πλαστικά είναι στην πρώτη θέση. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στα πλαστικά στη θάλασσα, αλλά και τα πλαστικά στη φύση και στην ύπεθρο. Και λυπάμαι που εστιάζουμε τόσο πολύ στα πλαστικά στη θάλασσα. Υπάρχουν και μικροπλαστικά τα οποία εμφανίζονται και στα τρόφιμα, διότι ε, τα βρίσκουμε και στα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές ε, και αλλού. Και επίσης, ε, θα ήθελα να πω κάτι για τα φρικτά οξοπλαστικά. Ε, θα ήθελα να υπάρχει κάτι ακόμα γι' αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι παγιωμένη η θέση μας. Ε, συμφωνώ και με κάποια που είπαν οι συνάδελφοι και η κυρία Ρης ε, για τα φίλτρα και τις γόπες των τσιγάρων. Ε, το βρίσκω επονίδιστο ότι εξακολουθεί να είναι πρόβλημα το συγκεκριμένο θέμα. Το κάπνισμα είναι ε, πρόβλημα από μόνο του ούτως ή άλλως. Τα φίλτρα και οι γόπες λοιπόν είναι πρόβλημα διότι βρίσκονται στη φύση πεταμένα παντού. Θα ήθελα λοιπόν κάτι για αυτή την πρόταση και χαίρομαι ε, που ασχολούμαστε και με τις ελαφρές παραστικές ε, σακούλες. Ε, όταν έκανα την πρότασή μου χρειάστηκε να το δεχτώ διότι δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί, αλλά χαίρομαι που πλέον βρήκαμε έναν τρόπο να το συμπεριλάβουμε στο όλο ζήτημα. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο συζητούσαμε ήταν τα επικίνδυνα χημικά στα πλαστικά. Αν θέλουν να ξανά χρησιμοποιούνται τα πλαστικά και να ανακυκλώνονται κατά θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνονται, ποια είναι η χημική σύσταση αυτών των πλαστικών. Τώρα μας λέτε ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλες τις ουσίες ε, που περιλαμβάνονται στην νομοθεσία REACH, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένα ε, σχέδιο για την επισήμανση. Ε, και είναι καλό το ότι θέλουμε να προχωρήσουμε για αυτό το θέμα. Ο, όσον αφορά την αρχή ο πληρώνει, ούτως ή άλλως ήδη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εδώ και υπάρχει και μεγάλη εφηβρωτικότητα. Ε, ο κόσμος βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε αυτή την ευθύνη και αυτή τη στιγμή κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να καταβάλει κάποιο πρόστιμο ή θα υποχρεωτηθεί να πληρώσει, Συνήθω γίνεται πιο καινοτόμο και πιο εφεύρετικό. Ε, Κυρίω για του παραγωγού, και ίσω θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή την πτυχή γιατί είναι σημαντική. Ποσοτικές μειώσει και στόχοι και τα όσα προτείνει η κυρία Ρης ε, και τις, ε, ε, θα επιβληθούν στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση αυτής της πτυχής. Και όσον αφορά ε, συσκευασίες τροφίμων, είναι καλό μεν που προτείνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ε, χαρτόνι ανταυτού, διότι ε, θα πίνει κανείς ε, ένα χυμό μέσα από χαρτόνι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πλαστικό. Ε, και πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Είναι πολύ πιο ευχάριστο το γεύμα σου να φέρεις ένα πιάτο, να το πλύνεις μετά. θα μπορούσε κανείς να το εξετάσει και αυτό ως εναλλακτική λύση. Χρειαζόμαστε αξιολόγηση επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας αναφέρει το στόχο της μείωσης ε, κατά 70 ε, με 80%. Ε, είναι πολύ καλός ο στόχος αυτός και καλό θα ήταν να το θέσουμε αυτό το στόχο. Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ρής και τους άλλους εισηγητές και εσκαιώδεις εισηγητές ή μάλλον να τους ζητήσω να έχουν κατά νου ότι ε, η ε, μείωση των αποβλήτων είναι πρώτη προτεραιότητα. Και μετά έχουμε την επαναχρησιμοποίηση. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά την πρόληψη όμως πρώτα, γιατί πάντα προτιμούμε την πρόληψη. Ε, πλαστικά μιας χρήσης. Μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με βιοδιασπόμενα πλαστικά, αλλά αυτό δεν είναι κατάλληλη πρόληψη και δεν αρκεί, διότι εξακολουθεί να έχει κάποιες ουσίες στο διασπόμενο πλαστικό που είναι επιζήμιες για τη φύση. Να βρούμε λοιπόν έξυπνες λύσεις για να αποφύγουμε τα πλαστικά μιας χρήσης. Και τέλος να σας πω ότι ένα μικρό νησί στη Δανία, το Φέινερ, δεν μπορεί να το γνωρίζετε κάποιοι από εσά, ε, απαγόρευσε τα μπαλόνια. Γιατί στις ακτές τους προς τα δυτικά είναι γεμάτο με μπαλόνια και μάλιστα φτάνουν λέει από την Αγγλία με τους δυτικούς ανέμους ε, ε, διασχίζουν τη Βόρεια Θάλασσα και καταλήγουν στις παραλίες τους. Ε, επομένως, οι, άνεμοι αυτοί δεν θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι λοιπόν θα υπάρχει επιβάρυνση ακόμα και μετά τον Brexit. Ε, αυτά ευχαριστώ πολύ κύριε Αρίς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γι' αυτό και υπάρχει μεγάλος κατάλογος ομιλητών. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε ένα όριο χρονικό στις παρεμβάσεις σας. Κύριο Πιεντετσίνη, τελευταίο σκιώδη. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσουμε να μειώνουμε του χρόνου ε, παρέμβαση από τον επόμενο. Ε, γιατί εγώ είμαι σκιώδη ηγητή, επομένω πρέπει να έχω χρόνο. Είναι σαφές λοιπόν για όλους ότι υπάρχει μια παγκόσμια περιβαλλοντική ε, ανάγκη, διότι πρέπει να μειώσουμε την ε, ε, κατανάλωση πλαστικών, το γνωρίζουν αυτό όλοι οι πολίτες, αλλά και επίσης διότι βλέποντας τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν μεγάλα μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ε, και ε, να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας ε, για τους πολίτες. Εμείς συμφωνούμε με την εισηγήτρια, την κυρία Ρή, την οποία ευχαριστούμε για τα όσα έκανε μέχρι τώρα, κυρίως όταν αφορά για στόχους μείωσης για τις βόπες των τσιγάρων που είναι από πλαστικό καθώς επίσης και για τις ε, πολύ ελαφριές πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα αντικατασταθούν από ε, σακούλες τις οποίες μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε, για να συμφωνήσω και με την κυρία Άουκεν. Και επίσης για λόγους υγιεινής θα μπορούσαν ίσως να αντικατασταθούν και από βιοδια... βιοδιασπόμενο ε, προϊόντα. Όσον αφορά τα απόβλητα, ναι, θα πρέπει να υπάρχει εκτεταμένη ευθύνη, αλλά δεν θα πρέπει ε, να ξεχνούμε ότι όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη των παραγωγών, αλλά και από τους πολίτες, ο οποίος θα πρέπει και αυτό ή να κάνουν κάτι για να υπάρχει μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα και λιγότερα απόβλητα. Θα πρέπει ε, να προβλέπονται κυρώσεις, για παράδειγμα, για όσους πετάνε ε, σκουπίδια σε δημοσίους χώρους και να επιβραβεύονται κάποιοι οι οποίοι σκοπεύουν ε, ή φροντίζουν να καθαρίσουν για παράδειγμα ακτές. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι ο στόχος της μείωσης, το είπε τώρα η κυρία Όκεν, και επίσης ε, να καθαρισουν για παραδειγμα κτες ο βασικος στοχος θα πρεπει να ειναι ο στοχος της μειωσης το ειπε τωρα η κυρια οκεν και επισης να χρησιμοποιουνται άλλες δυνατότητες αντί για μπουκάλια πλαστικού. Ε, η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του 50%. Το λέω στην εισηγήτρια γιατί έχουμε στοιχεία που μας επιβεβαιώνουν ότι αυτοί οι στόχοι είναι ρεολιστικοί και μπορούμε να τους επιτύχουμε. Δεν είναι σαφής η λόγοι για τους οποίους η εισηγήτρια αποκλεί τα ανθρακούχα ποτά ε, από αυτά τα οποία θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται άλλες συσκευασίες, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και επίσης θα πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός για το τι είναι βιοδιασπόμενο και τι ε, είναι κομποστοποίηση. Και εδώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Παολίτσι. Αν για ιατρικούς σκοπούς και για λόγους ασφαλείας στα νοσοκομεία είναι απαραίτητο, θα μπορούσε ίσως να υπάρχει μια παρέκκληση για τα πλαστικά μιας, είδης, ε, μιας χρήσης, αλλά μόνο για βιοδιασπόμενα πλαστικά. Ε, να πω ότι για μας δεν υπάρχει κανένα νόημα ε, να λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τη χρήση πλαστικών συσκευασιών εάν δεν ορίζεται επακριβώς το όρος ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία, ένα σαφής αριθμητικό στόχος, τον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μέσω ε, ε, ε, συστημάτων χρήσης, πρόληψης και επίσης μας ενδιαφέρει και το πεδίο εφαρμογή. Η πρόταση αφορά 10 προϊόντα πλαστικών μιας χρήσης που αποτελούν το 70% των αποβλήτων που βρίσκονται στι ακτέ μα. Επομένω έχουμε αρκετά δεκάδε εκατομμύρια τόνων αποβλήτων. Το να συμπεριλάβουμε στους καταλόγους και τα μπαλόνια. Ε, καταλαβαίνω αυτό που λέει η κυρία Άουκεν, αλλά και στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε 5 χιλιόγραμμα πλαστικού σε όλες τις ε, ε, ακτές και παραλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για πράγματα τα οποία έχουν διαφορετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και νομίζω ότι δεν θα πρέπει εδώ να υπερβάλλουμε, είναι μια υπερβολή που ε, μπορεί να θεωρηθεί και γελία σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος, όσον αφορά την έκκληση για την ανάγκη διαφάνειας και την παρουσία επικίνδυνων ουσιών για τα προϊόντα, πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται σωστά και να μπορούν να επιλέξουν ε, και να καταναλώνουν υπεύθυνα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. So, uh, Λοιπόν, κάθε παρέμβαση έως δύο λεπτά σας παρακαλώ, γιατί είναι πολύ μακροσκελής ο κατάλογος ομιλητών και έχουμε και άλλα τρία θέματα στην ημέρησια διάταξη, τα οποία επίσης θα απαιτήσουν χρόνο. Κύριος Ρο, που είναι εισηγητής ε, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Άγκρη. Δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, όπως είπατε, είμαι συντάξη γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής Γεωργίας, η οποία θα γνωμοδοτήσει στη δική σας Επιτροπή. Σήμερα το πρωί μάλιστα συζητήσαμε το θέμα αυτό και ήρθα εδώ για να ακούσω τη δική σας συζήτηση. Και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι η πλειονότητα των σχολείων που ακούστηκαν από όσους έλαβαν το λόγο ευθυγραμμίζονται και με τις δικές μας απόψεις. Θεωρώ ότι το έγγραφο που έχει προετοιμάσει η Κομισιόν είναι καλό, αποτελεί μια θετική βάση για τη συζήτηση που θα γίνει. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθεί το κείμενο αυτό, ώστε να μην χρειάζεται σε έξι μήνες να επανέλθουμε στο κείμενο αυτό με βελτιώσεις. Ας γίνουν τώρα. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι γιατι ως αφετηρία ως βάση. Είναι πολύ θετικό το κείμενο αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων, γιατί κάθε μέρα ακούμε και κάτι νέο όσον αφορά τη χρήση των πλαστικών. Για παράδειγμα, σήμερα, όταν πηγαίνει κανείς σε ένα κατάστημα, Μπορεί να δει ότι ένα λάχανο είναι συσκευασμένο μέσα σε πλαστική μεμβράνη, ενώ κάποιο άλλο λάχανο μπορεί να μην είναι συσκευασμένο σε μεμβράνη. Το ίδιο και με τα αγκούρια. Που πραγματικά είναι δυσνόητο. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς. Επίσης, πρόσφατα πήρα δώρο από, από ε, ένα, ένα χυμό που αγόρασα, ένα πλαστικό ποτήρι και ένα γυάλινο ποτήρι. Το πλαστικό ποτήρι ήταν ξανά συσκευασμένο σε μια άλλη πλαστική συσκευασία. Πέρσι εγώ διοργάνωσα ένα διαγωνισμό που προσήλκησε προσέλκυσε πολλούς νέους ανθρώπους και θέμα αυτού του διαγωνισμού ήταν τι θέλετε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα που έλαβε τις περισσότερες απαντήσεις ήταν ε, η μείωση των πλαστικών και η προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να δούμε πραγματικά την χρονική καταλληλότητα και των προτάσεων που υποβάλλουμε. Και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στα κείμενά μας να γίνεται αναφορά συστηματική και στα μικροπλαστικά, τα οποία αποτελούν υποπροϊόν της διάσπασης των πλαστικών ουσιών στη φύση και αυτές, αυτά τα μικροπλαστικά είναι και τα πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης χρησιμοποιούνται πλαστικά προϊόντα στη γεωργία τα οποία δεν συλλέγονται και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει και αυτό το θέμα. Όχι εις βάρος των γεωργών, αλλά εις βάρος των κατασκευαστών αυτών των προϊόντων. Σε δύο εβδομάδες, όπως ε, σας είπα, θα έχουμε ολοκληρώσει και τη σύνταξη της και θα την έχετε στη διάθεση σας. Κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία ρή διότι αύξησε το επίπεδο φιλοδοξία τη πρόταση στο σχέδιο εκθεσή τη. Επίση, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε την υπόσχεσή τη να προτείνει ε, σύντομα μία νομοθετική πρόταση, διότι ε, υπάρχει μία επίγουσα ανάγκη, η οποία γίνεται όλο ένα και πιο επίγουσα. Η ρήπανση από πλαστικά και κυρίω ε, η ρήπανση από πλαστικά στι θάλασσε και είναι μια πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με δράσεις όσο το δυνατόν πιο μετριασμένες μεν, αλλά και πιο αποτελεσματικές επιτρέψτε μου να πω. Από πλευράς λοιπόν αποτελεσματικότητας των προτάσεων, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αντίστοιχη με αυτό το οποίο υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οδηγία για τις πλαστικές σακούλες, την οποία συζητήσαμε ε, αναλυτικότατα και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα από την απαχώρευση της παραγωγής, μέτρα ευαισθητοποίησης, ε, μέτρα μείωσης της κατανάλωσης, αλλά και την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού. Και αυτό απέδειξε στην πράξη ότι μπορούμε να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και έχουμε μια ουσιαστική μείωση της πλαστικής σακούλας τα τελευταία χρόνια. Ε, ναι, με λοιπόν αφήνουμε στην άκρη τη μέθοδο. Θα ήθελα να προτείνω και κάτι ε, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επίκριση. Ε, τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά, δηλαδή πιο αυστηρά για τα πλαστικά τα οποία επηρεάζουν περισσότερο τις ακτές μας ε, και τα βλέπουμε περισσότερο στις παραλίες και τις ακτές. Θεωρώ ότι είναι μια αρχή η οποία είναι δίκαιη και θα ολοκληρώσω με το εξής πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχουν αμφισημίες στην νομοθεσία, ε, διότι θα οδηγήσουμε σε σύγχυση ε, μεταξύ αυτής της οδηγίας ε, και κάποιες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, όπως την οδηγία για τα παιχνίδια ή την οδηγία για τη συσκευασία, η οποία μόλις αναθεωρήθηκε στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις της ε, ανακύκλωσης ε, και της ανακύκλωσης ε, της διαχωρισμένης, θα πρέπει εδώ να έχουμε εκτεταμένη ευθύνη των παραγωγών. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ποιότητα της εργασίας της και την Κομισιόν για το φιλόδεξο χαρακτήρα της πρότασης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, διότι βρισκόμαστε σε μια τραγική κατάσταση. Σας υπενθυμίζω μερικούς αριθμούς. Μέχρι σήμερα, 10 δισεκατομμύρια τόνοι ε, παραγωγής πλαστικών και η μισή ποσότητα καταλήγει στη φύση και στο βυθό των ωκεανών αλλά θα πρέπει να έχουμε ε, επίσης υπόψη και τον αριθμό αύξησης του πληθυσμού. Ο πληθυσμός θα είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια κατοίκους το 2100 και μέχρι το 2050, αν εξακολουθήσουμε με τον ίδιο ρυθμό παραγωγής πλαστικών, θα πρέπει να δούμε ότι θα υπάρξει μία πρόοδος 28,5 δισεκατομμυρίων τόνων μέχρι το 2050 περισσότερο από όσο η ανθρωπότητα παρήγε και κατανάλωσε ως σε πλαστικά μέχρι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα που να μην είναι ημίμετρα. Και πολλοί το τόνισαν, νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε ε, τα πλαστικά μιας χρήσης. Δεύτερον, όσον αφορά τα φίλτρα των τσιγάρων. Είναι πραγματική μάστιγα. Πάνω από τρία δισεκατομμύρια γόπες καταλήγουν στη φύση. Πρέπει να τις απαγορεύσουμε. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί απέναντι ε, στους καπνοπαραγωγούς ε, και πάρα πολλά άτομα ξέρουν ότι καπνίζουν πλαστικά ε, και ότι αυτό το υλικό θα καταλήξει στο βυθό της θάλασσας. Η ε, βιομηχανία του καπνού που είναι από τις πιο ρηπογόνες είναι η μόνη που δεν έλαβε κανένα μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι εφόσον πρόκειται για το θέμα της ευθύνη. Υπάρχει βεβαίως μια ευθύνη των καταναλωτών. Βεβαίως πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά δεν θα πρέπει να μετακυλήσουμε ε, την ε, ευθύνη στους καταναλωτές και να αφήσουμε κατά μέρο τους παραγωγούς, διότι η παραγωγή είναι υπεύθυνη. Ο Κύριε Γραμματικάκης έχει το λόγο. Έχω τον παρελθόν, κυρία Πρόεδρε, ότι η ρήπανση των θαλασσών από έχει περάσει ένα κρίσιμο όριο και συνεπώς θα πρέπει να είμαστε τολμηροί στις λύσεις που προκρίνουμε. Και αυτό ακόμα και αν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποιες από τις αγαπημένες μας συνήθειες. Η σχετική πρόταση της Επιτροπής αποτελεί αναφυσβήτα ένα θετικό βήμα και βελτιώθηκε πάρα πολύ από τις προτάσεις της συγγήτριας. Φοβούμε όμως ότι ακόμα δεν είναι αρκετά τολμηροί. Έτσι, ενώ πολλές καλές ιδέες έχουν προταθεί, είναι δυστυχώς πολύ δύσκολο να υπολογίσει κανείς την αποτελεσματικότητά τους. Για παράδειγμα, η πρόταση ζητά τη σημαντική μείωση κατανάλωσης για δοχεία ή κουτιά. Τι σημαίνει όμως σημαντική μείωση, μπορεί ένα 10% να θεωρηθεί σημαντική μείωση, ένα 20%, ένα 30%. Είναι αυτό αρκετό. Και γιατί δεν προσθέτουμε και άλλα προϊόντα στον ίδιο στόχο, νομίζω ότι επιβάλλεται να δούμε πιο προσεκτικά ποια προϊόντα μπορούν να υπαχθούν σε μια πιο αυστηρή ρύθμιση. Επίσης, θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας. Ο στόχος μείωσης της κατανάλωσης πρέπει να επιτευχθεί έξι χρόνια μετά την εσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή σε 8 ή 9 χρόνια από σήμερα, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Το ίδιο ισχύει και για την αξιολόγηση της οδηγίας που είναι απαραίτητη για να κρίνουμε εγκαίρως την αποτελεσματικότητά της. Συμπερασματικά, το πρόβλημα της ρήπασης των θαλασσών, αγαπητοί συνάδελφοι, το είπατε οι περισσότεροι που μιλήσατε, είναι επίγον και η κρισιμότητά του διαρκώς οξύνεται και είναι επίγον για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη χώρα μου που είναι πρικισμένη με μεγάλη έκταση ακτών. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί στην πηγή του και δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να χάσουμε μια ακόμα ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Ντόφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος ε, γιατί τη μείωση των πλαστικών βεβαίως μας ενώνει όλους. Αλλά ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους κλίμακα. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ή δημιουργείται εντύπωση από αυτά που ακούμε ότι εμείς με μια ευρωπαϊκή στρατηγική μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την τεράστια ε, κοιλίδα πλαστικών που υπάρχει στον Ειρηνικό ωκεανό ή στη διόρυγα του Παναμά. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Πάνω από το 90% των πλαστικών στις θάλασσες προέρχονται από 10 ε, ποταμούς. 8 από αυτούς στην Ασία και 2 από αυτούς στην Αφρική. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και να τη συνεκτιμούμε. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι πρόκειται και για ένα θέμα ανακύκλωσης και ορθής λειτουργίας της κυκλικής οικονομίας, διότι ακόμα και τα βιοδιασπόμενα πλαστικά δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον, ακόμη και αν βιοδιασπώνται τα υλικά αυτά μετά από πολλά πολλά χρόνια. Κανένα είδο αποβλήτων δεν πρέπει να καταλήγει στο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει στο πλαίσιο μια κυκλική οικονομία να επαναχρησιμοποιείται και να ανακυκλώνεται. Βεβαίω, τα καπάκια μπορεί κανείς να τα κατασκευάζει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάνονται από το, από μπουκάλι, να μένουν πάνω. Το έχουμε δει σε κονσέρβες εδώ και πολλά χρόνια. Το ανοιχτήρι, το δαχτυλίδι μένει πάνω στο καπάκι. Δεν το ξεκολλάς, οπότε δεν καταλήγει στο περιβάλλον. Μην καταλήξουμε όμως και σε ακρότητε να απαγορεύσουμε τώρα τα μπαλόνια από τα παιδάκια έχοντας την ψευδέστηση ότι έτσι θα σώσουμε το περιβάλλον. Α δούμε τα πράγματα στη σωστή του κλίμακα, ας κάνουμε αυτά που πραγματικά θα αποφέρουν αποτελέσματα και όλα τα άλλα α τα αφήσουμε κατά μέρο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Σπότ paní Jenom Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατεπηγόντως. Ε, και είναι και το μόνο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, διότι πουθενά δεν βρήκα ε, τι γίνεται συγγνώμη που το λέω τώρα, τι γίνεται λοιπόν με τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων. Πρόκειται για μικροστοιχεία, από νάνο έως μικροστοιχεία ε, και υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ούτε καν αυτοί που οι οποίοι παράγουν ελαστικά οχημάτων δεν μπορούν να μας πούνε ποια είναι αυτά τα μικροσωματόδια ε, τα οποία περιλαμβάνονται στα ελαστικά ε, πρόκειται για πλαστικά τα οποία επηρεάζουν την υγεία μας και εδώ στην Ευρώπη. Δεν είναι θέμα για τους ωκεανούς, είναι κάτι το οποίο πραγματικά ε, ε επηρεάζει την δημόσια υγεία. Και είναι και κάτι το οποίο δεν έχει σκεφτεί κανείς στην Ευρώπη μέχρι τώρα ούτε ο κλάδο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη νομοθεσία θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και το θέμα αυτό, να υποβάλουμε και κάποιε τροπολογίε. Έχω ετοιμάσει εγώ σχετικέ τροπολογίε και θα ήθελα να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει κατά πόσον θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και με αυτό το πρόβλημα εδώ στα πλαίσια αυτή τη οδηγία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα αποφύγω να επαναλάβω αυτά που είπαν προηγουμένω οι συνάδελφοι, διότι θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν έχει συζητηθεί επαρκώ ε, στην πρόταση οδηγία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε θα είναι οι συνέπειες ε, της απαγόρευσης των πλαστικών μιας χρήσης. Η ρήπανση από πλαστικά είναι μία από τις μεγαλύτερες επίγουσε ανάγκες, τις οποίες θα πρέπει να παρέμβουμε με αποφασιστικότητα και με σαφήνεια. Επομένω, είναι ευπρόσδεκτα τα μέτρα επανόρθωση, μεν, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μακρόπνοα, διότι με αυτέ τι οδηγίε ουσιαστικά καθορίζουμε το νέο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και προσδίδουμε μορφή στα νέα μοντέλα βιωσιμότητας του πλανήτη. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στις συλλογικέ συμπεριφορές και να δούμε και τι εναλλακτικά υλικά έχουμε στη διάθεσή μας. Δηλαδή, πώς θα κατευθυνθεί η αγορά την επομένη της απαγόρευσης. Από κάποιες έρευνες τις οποίες διάβασα φέτος το καλοκαίρι, διαπίστωσα ότι υπάρχουν δύο άμεσες εναλλακτικές λύσεις για τα ε, πιάτα και τα ποτήρια, τα πλαστικά τα βιοπλαστικά και ο πολτό, ε, τα οποία όμως ε, κυρίως ε, προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγή βιοπλαστικών αυτή τη στιγμή είναι γελία σε σχέση με αυτά τα οποία χρειάζεται η αγορά και δεν επιτρέπουν να γίνει αντακατάσταση 100% των πλαστικών. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Πολλό δε μάλλον που το κόστος των βιοπλαστικών είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό της, του πολιτού που θα καταλάβουμε μεγάλο χώρο στην αγορά. Πολτό ο οποίος έχει δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχάς είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος από τα πλαστικά ε, πιάτα για παραγωγή πολτού η ενεργειακή κατανάλωση είναι ε, εντυπωσιακή επομένως το ε, αποτύπωμα του άνθρακα είναι πολύ μεγαλύτερο και επίσης υπάρχουν πολλά λειτουργικά προσκόμματα η πρώτη ύλη θα πρέπει να μεταποιηθεί κατά τρόπο νόστο, να επιτρέπεται η κομποστοποίηση και θα δημιουργείται ρήπανση, Απλώ θα είναι διαφορετική. Θα είναι αόρατη αυτή η ρήπανση, αλλά θα είναι εξίσου επιζήμια. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, να δούμε ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συλλογική συμπεριφορά των ανθρώπων και επίσης να ξέρουμε ότι στη φύση θα έχουμε βιοπλαστικό και πολτό τα οποία έχουν μικρότερους χρόνους ε, μεν ε, ρήπανσης αλλά θα συνεχίσουν να ρηπαίνουν τι θάλασσές μας. Ευχαριστώ κυρία Ντάλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια και βεβαίως ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα και την πρόληψη ε, και να δούμε τις υποδομές, την ε, παραγωγή και βεβαίως την εφαρμογή. Θα ήθελα να συγχαρώ την, την εισηγήτρια που ενισχύει την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την μείωση. Βεβαίως θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές και οι καταναλωτές να ασχοληθούν. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται, να αλλάξουν την συμπεριφορά τους, να ευαισθητοποιούνται, αλλά και η παραγωγή επίσης για την χρήση, την βιώσιμη των προϊόντων. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των πολιτών μας και το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε μεθοδολογία αποτελεσματική που θα επιτρέψει συγκεκριμένα μέτρα στο επίπεδο των κρατών μελών και στην εφαρμογή. Οι, τα, οι θα πρέπει να βελτιώσουν τις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και να ευαισθητοποιήσουν τους παραγωγείς και τους καταναλωτές. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο κυκλικό μοντέλο θα πρέπει να έχουμε την ορολογία την κατάλληλη για να μην υπάρχει σύγχυση, να υπάρχουν οι κατάλληλοι ορισμοί για να μην έχουμε επιπτώσεις απρόβλεπτες ε, και θα πρέπει να έχουμε τον στόχο 90% για την συλλογή ε, και θα πρέπει τα μέσα να χρησιμοποιηθούν που πρότεινε η συγγήτρια θα πρέπει βεβαίως ο ορισμός της ε, ξεχωριστής συλλογής, της επιλεκτικής συλλογής να αναφέρεται εδώ. Θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο εργασίας ε, για την καλή εφαρμογή για ασφαλέστερο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Α, έχουμε κανέναν άλλον, καμιά άλλη παρέμβαση. Όχι. Ε, Κύριε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαίρετη εισήγηση ε, και η εισήγηση αυτή είναι ε, η αρχή ε, της, εδώ της εργασίας στο Κοινοβούλιο και για φιλόδοξο νομοθετικό έργο. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια για κάθε σημείο της εισήγησης αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά προκαταρκτικά. Διαβάσαμε την εισήγηση με ενδιαφέρον ε, και ακούσαμε και επίσης ε, τη γνώμη άλλων επιτροπών, Επιτροπή Γεωργίας ε, και θα ακούσουμε και άλλες επιτροπές τις επόμενες μέρες και χαιρόμεθα για την προσέγγιση η συζήτηση που είχατε σε αυτήν την Επιτροπή σχετικά για το πλαίσιο για, το, για την οδηγία, πλαίσιο για τα απορρίμματα, μιλήσατε για πρόληψη και νομίζω ότι αυτή η οδηγία αφορά κυρίως την πρόληψη. Σημειώσαμε στα μέτρα που πρότεινε η συγγήτρια μερικά μέτρα πιο φιλόδοξα από αυτά που προτείναμε εμείς ε, σχετικά με την ε, προθεσμία, ε, σχετικά με την ελάχιστο περιεχόμενο περιεκτών και ανακύκλωση, η σήμανση και διάφορα μέτρα να επεκταθούν οι υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών ε, και εκθέσεων το θέμα των φίλτρων. Το θέμα για τις σακούλες, τις πλαστικές, η εργασία μας είναι ε, συμπληρωματική με την, με την εργασία που γίνεται για την οδηγία σχετικά με τις συσκευασίες ε, σχετικά με τις σακούλες μεταφοράς ε, περιλαμβάνονται οι πολύ λεπτές σακούλες ε, και ίσως μπορεί να υπάρχει εξαίρεση εάν έχει επιτευχθεί ο συνολικός στόχος τα στοιχεία που έχουν ήδη ε, συλλεγεί για τις σακούλες δείχνουν ότι ο στόχος αυτός είναι αποτελεσματικό. σχετικά ε, με τον στόχο για την ανακύκλωση δεν υπήρχε στην πρόταση ε, της Κομισιόν διότι έχει τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις όπως και τα άλλα πλαστικά σχετικά με την επιλεκτική συλλογή για να έχουμε ε, κάτι το ξεχωριστό, είναι ένα σήμα αρκετά σημαντικό, ένα σημάδι, ένα μήνυμα, μια στρατηγική χρειάζεται και θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ε, στην οδηγία σχετικά με τις συσκευασίες, με τη συσκευασία γενικά και όχι να ασχοληθούμε μόνο με τα αντικείμενα μιας χρήσεως. Υπήρξε μια εκστρατεία η οποία επεκτάθηκε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ε, ούτω ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δούνε ποια δέσμευση μπορούν να αναλάβουν ε, σχετικά με τα προϊόντα τους και ελπίζουμε ε, να δούμε μετά τι περαιτέρω μέτρα θα ήταν αναγκαία. Σχετικά με τον εξοπλισμό αλληλείας δεν ήμασταν σε θέση να υποστηρίξουμε αυτόν τον στόχο διότι πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία και τα δεδομένα, αλλά πρέπει να πω ότι ο στόχος ανακύκλωσης θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω κίνητρο για τους παραγωγούς, ούτως ώστε να λάβουν μέτρα για την ανακύκλωση των αλλιευτικών εργαλείων. Υπάρχουν δυνατότητες που και μπορούμε να έχουμε προσεγγίσεις πιο κυκλικές και είναι το μήνυμα το οποίο εκφέρει στην κοινότητα την αλλιευτική ή κομισιό. Αλλά βεβαίως πρέπει να ξέρουμε πόσα ανακτώνται, πόσα, ε, πόσα από αυτά τα εργαλεία, τα υλικά επιστρέφονται στις ακτές ανακτώνται κατά κάποιο τρόπο. Λυπούμαστε για μερικές τροπολογίες που περιορίζουν ε, την ορισμένα μέτρα υφορίας σχετικά με τις απαιτήσει ε, σχεδιασμού. Η πρόταση της Κομισιόν βλέπει ε, πώς ασχολούμεθα με τα θαλάσσια απορρίμματα ε, και με τα απόβλητα και αυτό περιλήφθηκε στην οδηγία που ζητάει από την να καθαρίζουν τις ακτές ε, τα, τα κράτη και διότι οι καταναλωτές είναι η βασική ε, πηγή αυτών των απορριμμάτων. Αλλά συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός ούτως ώστε να υπάρχει αναλογικότητα για τον λόγο αυτό αντί να εξετάζουμε την πλήρη εξαίρεση για τους ε, ποταμούς ε, από ευθύνη θα πρέπει να επιζητήσουμε μια ισορροπία ε, σχετικά με τα καλύματα, με τα καπάκια των διαφόρων ποτών βεβαίως ε, η συγγήτρια θέλει να εξαιρέσει αυτά τα προϊόντα. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για το θέμα αυτό διότι βλέπουμε πάρα πολλές φιάλες, φιάλες στο τραπέζι μας με μπλε καπάκια, με κόκκινα καπάκια. Τι δηλαδή, με τα μπλε καπάκια θα απαγορεύονται και με τα κόκκινα καπάκια θα εξαιρούνται, πώς θα γίνει αυτό για να μειώσουμε την ζημία στο περιβάλλον. έχουμε πλήρη συνείδηση των θεμάτων που απασχολούν την βιομηχανία, τους παραγωγούς ποτών και είμαστε διαθέσιμοι για να βρούμε έναν καλό τρόπο για να υπάρξουν οι κατάλληλες αλλαγές και παρακολουθήσαμε τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι ορισμοί και ε, διευκρινήσεις σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από αυτήν την οδηγία. Ε, οι περιέκτες τροφίμων ε, και εναλλακτικέ λύσεις πρέπει να υπάρχουν για το θέμα αυτό. Η Κομισιό είναι διατεθειμένη να δώσει καλύτερη ερμηνεία και σαφήνεια, ούτως ώστε να διευκολυνθεί το εθνικό επίπεδο Επίσης έχουμε προϊόντα πλαστικά τα οποία απορρίπτονται στο περιβάλλον που δεν είναι τελείως πλαστικά αλλά που δημιουργούν την ίδια ζημία. Χρειάζεται λοιπόν εδώ σαφήνεια. Και τελευταίο σημείο υπήρχε ένα θέμα που τέθηκε από την κυρία Ντεμεσμάκερ σχετικά με την μείωση Βεβαίως δεν έχουμε την βασική γραμμή και στοιχεία. Ας εξετάσουμε πρώτα την, το θέμα της μείωσης. Ο αριθμός χρήσεων αν θα αυξηθεί σημαντικά αν δεν κάνουμε κάτι. Η μείωση αυτή καθεαυτή είναι κάτι που θα πιέζει τα κράτη-μέλη να δράσουν. Να δούμε πόσο σημαντική μπορεί να υπάρξει μείωση με αυτήν την οδηγία και όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα, τους αριθμούς, τα στοιχεία που θα μπορούμε να περάσουμε σε συγκεκριμένο στόχο. Από τον κύριο Πότσο ένα σημείο ε, σχετικά με τα μικροπλαστικά που είναι ένα μεγάλο θέμα. κυρίως για τα ελαστικά, ε, για τα λάστιχα ε, θέμα των μικροπλαστικών είναι θέμα επεξεργασίας. Αν υπάρχουν ε, πλαστικά θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ε, στα ελαστικά για να ξέρουμε αν περιλαμβάνονται τέτοια σωματίδια. Κόκκι. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρής και σας κυρία Πρόεδρε που οργανώσατε αυτήν την συζήτηση για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και για την εισήγηση αυτή ε, ε, η οποία χρήζει περαιτέρω διαπραγμάτευσης. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία ρίς Σας παρακαλώ όμως ε, εντός πέντε λεπτών σας παρακαλώ. Βεβαίως όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι αδύνατο να απαντήσω σε όλους. Ο κύριος Φλόρενς είχε δίκιο που είπε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή την οποία έχουμε αυτή την στιγμή ε, και ε, η Κομισιό ε, θέλει στοιχεία θετικά αναφέρθηκε κάτι από έναν παππού για τα εγγόνια του. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις ε, για τα μπαλόνια, αν θέλετε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Βεβαίω, έχουμε μια εναλλακτική λύση, η οποία είναι εύκολα διαθέσιμη. Βεβαίω, δεν θέλουμε να εξαλείψουμε τη χαρά των ε, παιδιών. Το... Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο τα ε, ε, επικίνδυνες ουσίες. Θα δούμε πώς θα συνεργαστούμε μαζί για να ενοποιήσουμε το κείμενο. Οι εξαιρέσεις βεβαίως αναφέρονται αναφέρονται από την Κομισιόν στην πρόταση. Ο κύριος Ντεμεσμακέρ νομίζω ότι είπατε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ, διότι έχουμε πλήρη συνείδηση ε, της Κατάσταση έχουμε τις γνωμοδοτήσεις. Δεν έχουμε κάθε φορά τέτοιες γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις ανησυχίες. Έχουμε την ανθεκτικότητα ε, των υλικών αυτών. Έχουμε την ευκαιρία στη ζωή μας ε, και όλοι οι εμπειρογνώμενες μας λένε ότι πρέπει να υποφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία εδώ και τώρα, κύριε Ντάρμαν, ε, σε μια ανταλλαγή απόψεων αναφέρθηκε αυτό το θέμα το οποίο είπατε εσείς άρχισα προκαταρκτικά λέγοντας ότι δεν είναι γι' αυτό ότι δεν πρέπει να, η Ευρώπη να δράσει όπως έχει γίνει και με την, την κλιματική αλλαγή. Βεβαίως έχουμε συμβολή στην ρήπανση Ακούσαμε την απάντηση της Κομισιόν. Είχα την ίδια ανησυχία σχετικά με τα μικροπλαστικά. Επίσης τα συνθετικά, κλωστοϊφαντουργικά που έχουν ρήπανση μικροπλαστική είναι βεβαίως δύο θέματα, αλλά το προβληματισμός είναι κυρίως να δούμε αν είναι ε, το καλύτερο εδώ κείμενο ε, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ακολουθώ το δρόμο της Κομισιό. Ό,τι θα κάνουμε μαζί και δεν μίλησα για το θέμα των ορισμών ο κύριος Φεντουτσίνη η επάντηση της Επιτροπής. Έχουμε η παραγωγή μας λένε ότι δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν. Εγώ είναι δύσκολο να τους πούμε τι θα επιβάλλουν. Εγώ θέλω να στοιχηματίσω πάνω στην καινοτομία για το μέλλον Ακούσαμε αυτές τις ανησυχίες. Ε, είδαμε ότι η Κομισιόν αποδίδει σημασία στην ανακύκλωση, το 15% δεν είναι πολύ. Έχουμε βεβαίως τα ποτάμια που μας φέρνουν 85%. Στο 15% βεβαίως δεν ξέρω αν είναι φυκτό. Είναι ένα μίνιμουμ Κυρία Πρόεδρε, είμαι 20 χρόνια ε, εδώ Ευρωβουλευτής. Δεν είδα ποτέ τέτοια όθηση ε, θετική. Έχουμε το καλό timing, τον καλό χρονισμό ε, και έχουμε πάρα πολλές απόψεις θετικές. Βεβαίως θα υπάρξουν διχογνωμίες, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε και πίεση χρόνου. Αρχίζουμε με την επόμενη σύνοδο ε, του Στρασβούργου ε, για να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα πριν από τις εκλογές. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρίς και όλους τους άλλους συναδέλφους. Προθεσμία για τι ε, τροπολογίε είναι 4 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία θα γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, επίσης πολύ ενδιαφέρον, πρότυπα επιδόσεων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για νέα βαρέα οχήματα. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης που έχει συντάξει ο κύριος Eichhout. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να περιμένουμε ίσως μέχρι το λόμπι των μπαλονιών να εγκαταλείψει την αίθουσα. But I can recommend everyone to stay over because it's, uh, this, this topic is also very important. Αν και θα συνιστούσα σε όλους να μείνουν, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για τα βαρέα οχήματα. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα βαρέα οχήματα. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν εξετάσετε τη συμφωνία του Παρισιού, την οποία έχουμε υπογράψει όλοι, και το τι επιπτώσεις έχει όσον αφορά τους στόχους μας που επίσης έχουν ε, εγκριθεί από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για τις ε, μεταφορές χαμηλών εκπομπών, το συμπέρασμα είναι ότι ο κλάδος των μεταφορών θα πρέπει έως το 2050 να κινείται σε σχεδόν μηδενικές τιμές εκπομπών, ενώ ταυτόχρονα ο κλάδος αυτός είναι ο μόνος ο οποίος αυξάνει τις εκπομπές του Περίπου το 1 τέταρτο των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα προέρχονται από τον κλάδο των μεταφορών. Είναι ένα τομέα λοιπόν στον οποίο πρέπει να αναλυφθεί η δράση. Επίση γνωρίζουμε ότι οι μεταφορέ δεν ε, εντάσσονται στο ETS, εντάσσονται στο μηχανισμό επιμερισμού προσπαθειών και υπάρχουν μόνο εθνικοί στόχοι. πλέον τα πλέον κοστοαποδοτικά μέτρα λοιπόν ε, κινούνται στον τομέα των μεταφορών και ιδίως αφορούν τα νέα βαρέα οχήματα. Και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα και να εξασφαλίσουμε ότι ο κλάδος θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών δίνοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα κίνητρα για καινοτόμε λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν έως το 2050 σε μηδενισμό των, των εκπομπών. Αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό, σε 32 χρόνια θα πρέπει από σήμερα να θεσπιστούν τα κατάλληλα κίνητρα. Γι' αυτό και μας χαροποιεί η πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν δημοσιεύτηκε στα τέλη του Μαΐου και εμείς σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε μια διαδικασία fast track προκειμένου να κλείσουμε το φάκελο αυτό υπό Αυστριακή Προεδρία ακόμη. Πρόκειται για πολύ ε, φιλόδοξο στόχο, είναι πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν προθεσμίες υποβολής ε, τροπολογιών, έχω έρθει σε συνεννόηση με τους σκιώδεις, όμως συμφωνούμε όλοι, θα χρειαστεί να καταβλάλουμε όλοι μας προσπάθειες ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση η οποία θα εξασφαλίζει φιλόδοξους στόχους. Και έτσι τα πρότυπα και τα νέα βαρέα οχήματα θα συμβάλλουν στην αναγκαία αλλαγή στον κλάδο των μεταφορών με ορίζοντα τον εκμηδενισμό των εκπομπών. Εξετάσαμε λοιπόν τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν. Υπάρχει πάντοτε ανάγκη να διεξάγονται τέτοιες μελέτες αντικτύπου. Κάποιες φορές όμως έχω την αίσθηση ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν ακολουθεί την ίδια την αξιολόγηση που έκανε την μελέτη αντικτύπου που έκανε η ίδια η Κομισιόν. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχουσες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν στον κλάδο να μειώσει τις εκπομπές του ε, έως και 15 με 25% έως το 2025. Η Κομισιόν πάλι ε, αναφέρει ότι ο στόχος για τον, κλάδο, για τον έως το 2025 είναι το 15%. Μα αφού η ίδια η μελέτη που σας ε, αναφέρει ότι μπορεί να υπάρξει μείωση ακόμα και 20% με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, για ποιο λόγο να μην θέσουμε έναν τέτοιον ε, φιλόδοξο στόχο, αφού άλλωστε η, τα, η, τα καθαρά ωφέλη για την κοινωνία θα είναι τα μέγιστα με αν τεθεί στόχος 20%. Βεβαίω αυτό θα προκαλέσει υψηλότερο κόστο για του κατασκευαστέ. Αλλά νομίζω ότι ω νομοθέτε πρέπει να εξετάσουμε συνολικά τα κοινωνικά ωφέλη και αφού είναι εφικτό να επιτευχθούν αυτά τα ωφέλη, τότε νομίζω ότι πρέπει να τεθεί ο στόχος 20% για το 2025. Και επιπλέον, οι υπολογισμοί, υπολογισμοί αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη ε, οχημάτων μηδενικών εκπομπών παρά το γεγονός ότι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν ήδη ανακοινώσει και εξαγγείλει ότι έως το 2023-2025 ενδέχεται να βγάλουν στην αγορά ακόμη και τέτοια ηλεκτροκίνητα φορτηγά μηδενικών εκπομπών. Άρα ο στόχος είναι πέρα και από εφικτός. Μακροπρόθεσμα νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται για να καταλήξουμε στις μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Πρέπει να μπει ένας στόχος και για το 2030. Εκεί ο στόχος που έχει μπει είναι 45%. Ε, Βεβαίως υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά ζητήματα και γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί και ενδιάμεση αναθεώρηση. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι σε εκείνη την αναθεώρηση μπορεί να αλλάξει ο στόχος αυτός για το 2030, αλλά θέλουμε η αλλαγή, όποια αλλαγή γίνει στους στόχους, να είναι προς τα πάνω. Ακριβώς γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που πολύ πιθανό σε λίγα χρόνια μπορούμε ε, να επανέλθουμε ε, σε αυτούς τους στόχους που θέτουμε σήμερα και να πούμε «Μα γιατί ήμασταν τόσο μετριοπαθείς». Μείωση λοιπόν των εκπομπών είναι ένα από τα βασικότερα ζήματα που μας απασχολούν, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Πώς θα προωθήσουμε εκπομπές χαμηλές ή και μηδενικές. Πώς μπορούμε μάλιστα να καταλήξουμε και σε μια εντολή ΣΛΕΦ δηλαδή μηδενικές και χαμηλές εκπομπές. Κίνητρα για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Η μελέτη αντικτύπου αναφέρει ότι ένα κίνητρο δεσμευτικό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο σοβαρό ώστε ο κλάδος να επενδύσει στην έρευνα για την κατασκευή οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε ε, να ε, υπάρξει ρύθμιση νομοθετική για όλες τις κατηγορίες, γιατί αυτή τη στιγμή εντάσσονται μόνο ε, τέσσερις κατηγορίες στην πρόταση. Αντιθέτως με αυτό που προτείνουμε εμείς, ε, θα εξασφαλιστεί ότι η κατεύθυνση αυτή θα ακολουθηθεί σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τα λεωφορεία. Βεβαίως εντάσσονται στην πρόταση, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο μπροστά η τεχνολογία στα λεωφορεία, αν τα αφήσουμε εκτός εντολής, τότε θα ενδεχομένως να, να, να υπάρξει και μια επιβράδυνση στην εξέλιξη που υπάρχει. Γι' αυτό ενδεχομένως θα ήταν καλό να υπάρξει μια ξεχωριστή εντολή για τα λεωφορεία και τα, ιδίως τα υπεραστικά λεωφορεία. Μετά, κάποια ζητήματα που ενδεχομένω να μα απασχολήσουν στη διάρκεια των συζητήσεων. Προτείνουμε κάποια ευελιξία στη διάρκεια του χρόνου, ώστε αν οι κατασκευαστέ δεν καταφέρουν να επιτύχουν του στόχου του το 2025, θα πρέπει όμω να υπερβούν του στόχου για το 2030. Έτσι, η πρότασή μα του προσφέρει κάποια ευελιξία. Έχουμε διαγράψει το άρθρο 5 το οποίο ε, είναι και εκεί όπου η Κομισιόν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει αυτές τις υπερπιστώσεις ε, και την αξιοποίηση των μηδενικών ε, ε, εκπομπών οχημάτων. Θεωρούμε όμως ότι αυτός ο στόχος είναι αντιπαραγωγικός και γι' αυτό τον, τον διαγράψαμε. Επίσης ενισχύουμε κάποιες αρχές όπως αυτή που υπάρχει στα άρθρα 7 και κάναμε κάποιες, κάποιους σαφείς ορισμούς όσον αφορά τη διαφάνεια και τις δοκιμές. Γιατί από τα σκάνδαλα που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια ή ακόμη και χτε όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώ μετρούμε, τι ακριβώ συμβαίνει και πώ ακριβώ θα βελτιωθούν αυτοί οι ανεξάρτητοι έλεγχοι ώστε αυτά που μα υποβάλλουν ω στοιχεία οι κατασκευαστέ να ανταποκρίνονται, και στην πραγματικότητα. Τέλο, περιμένω κάποιοι να μιλήσουν και για αυτήν την, αυτό το τέλος ε, που ε, επιχειρεί να θεσπίσει η Κομισιόν. Ξέρω ότι σίγουρα θα τοποθετηθεί και η Κομισιόν, ωστόσο εγώ θέλω προκαταβολικά να εκφράσω την υποστήριξή μου σε αυτή την ιδέα της Κομισιόν, άλλωστε βασίζεται και στην ε, μελέτη αντικτύπου που η ίδια διεξήγαγε και θεωρώ ότι αυτό, αυτό που πρέπει να αποφευθεί είναι να μην βάλουμε τους κατασκευαστές απλά να πληρώσουν κάποια χρήματα και να τα αφαιρέσουν αυτά τα χρήματα από την έρευνα και την κοινοτομία. Να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στην έρευνα και την καινοτομία για την κατασκευή ε, οχημάτων χαμηλών και μηδονικών εκπομπών και όχι να δοθεί ε, κίνητρο στους κατασκευαστές να δώσουν απλά κάποια χρήματα, κάποιο τέλος για το γεγονός ότι κατασκευάζουν ρηπογόνα οχήματα και να ξεμπερδεύουν με αυτόν τον εύκολο τρόπο. Νομίζω όμως ότι παρόλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει, όλο και κάποιο συνάδελφος θα βρεθεί να το θέσει και θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έκχαουτ. Περνάμε στους κοιοδησίτες, αν είναι εδώ παρόντες. Ο κύριος Φιέλνερ καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Μπά για την εισαγωγή του. Καταρχάς να πω ότι εμένα με ανησυχεί το χρονοδιάγραμμα εν γέννη. Είναι πολύ αυστηρό ε, για νομοθεσία η οποία εισάγεται για πρώτη φορά. Δεν επικαιροποιούμε τίποτα. Είναι πρώτη φορά που υποβάλλεται τέτοια νομοθεσία και με ανησυχεί ε, το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να οδηγήσει σε κακή νομοθεσία, διότι πρέπει να έχουμε χρόνο να καταλήξουμε και σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Η μεγαλύτερη πρόκληση εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση, διότι πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι αυτό είναι το μέλλον και αυτή είναι η λύση ε, και ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για αυξημένη αποτελεσματικότητα των μηχανών εσωτερικής καύσης, οι οποίες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για αρκετό καιρό. δεν είμαι τόσο θετικά διακείμενος ε, ε, στην ε, πλήρη ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στη ζήτηση και ο λόγος είναι ότι κανένα από αυτά τα μεγάλα φορτηγά τα ηλεκτρικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα προκύψουν, υπάρχουν σχέδια για αυτά τα μεγάλα ηλεκτρικά φορτηγά, αλλά δεν έχει πουληθεί ούτε ένα μέχρι τώρα. Επομένως, το να λέμε ότι αυτή είναι η λύση και η μόνη λύση ε, νομίζω ότι είναι κάπως πρόημο. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πετύχουμε όλα τα υπόλοιπα ταυτόχρονα. Χρειαζόμαστε και υποδομέ, ε, νομίζω ότι υπάρχουν αναφορέ αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να κατασκευάζονται υποδομέ για υποστήριξη όλων αυτών και την παραγωγή ενέργειας, η οποία θα πρέπει να είναι και αυτή ε, ε, ε φιλική προς το περιβάλλον και σε ένα ρυθμό, που δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή και επομένω δεν είναι η λύση ε, προς το παρόν. Ε, σωστό είναι να δίνουμε κίνητρα. Εγώ όμως θα πήγαινα προς την αντίθεση σε σχέση με το μπας. Θα αύξανα το ποσοστό για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και θα ε, έβγαζα το όριο του 30%. Επίσης, η πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση εδώ δεν είναι αυτή με τους υψηλότερους στόχους ή την ε, με καλύτερη ζήτηση, αλλά να έχουμε απόλυτα σωστή ισορροπία μεταξύ των όσων κάνουμε εδώ, διότι αν αυτό το πρόβλημα είναι τόσο οξύ και τόσο μεγάλο όσο ισχυριζόμαστε, τότε δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν τα πάντα και να δίνονται ε, για οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε εδώ και τώρα και ταυτόχρονα να πιέζουμε για πράγματα για το μέλλον. Και εδώ έρχομαι στους στόχους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δύσκολο να επιτευχθεί μεν, αλλά μπορεί να ε, τα καταφέρουμε. Εξαρτάται πολύ από το πώς θα γίνει η αξιολόγηση της εκτίμησης επιπτώσεων. Και διαβάζοντα την εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή λέει 15% ε, μείωση το 2025 επιτρέπεται βάσει της παρούσας τεχνολογίας. Και επομένως γιατί δεν γίνεται αυτό. Και βλέπουμε ότι ε, τα λιπαντικά, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να οδηγήσει σε 4%. Ε, τα παραπετάσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τα ελαστικά ε, να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Εγώ περιμένω να το δω για να το πιστέψω. Περιμένω να δω τους υπολογισμούς ε, που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να κάνει αυτούς τους ισχυρισμούς. Διότι όταν εγώ συναντώ παραγωγούς ελαστικών λένε ότι η κατανάλωση είναι διπλάσια από αυτή που πιστεύουν ότι είναι τεχνικά ε, εφικτή ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο. Διότι είτε κάνουν λάθος και επομένως είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ή έχουν δίκιο και εγώ θα... Ε, παραιτηθώ και θα αρχίσω να πουλάω λιπαντικά, διότι εκεί είναι τα κέρδη στην αγορά. Μπορείς να έχεις 4% και... Α, έστω όμως ότι είναι σωστά. Ο στόχος του 2025 και πάλι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, διότι πολλές από τις εξελίξεις, τα λεωφορεία και τα φορτηγά τα οποία θα πολλούνται το 2025, σχεδιάζονται για τώρα. δεν προβλέπεται ένας νέος κινητήρας για το 2025. Ξέρουμε τι θα προκύψει και γνωρίζουμε περίπου το αποτέλεσμα. Μπορούμε να δούμε την κατανάλωση σήμερα για παράδειγμα και ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι Mercedes και η Scania κατά πάσα πιθανότητα θα τα καταφέρουν ενώ κάποιες άλλες, η Mandy, η Beko κλπ ε, θα τρέχουν από πίσω από τις εξελίξεις. Ξέρουμε, ένα-δυο θα χρεοκοπήσουν κιόλα. Αλλά αυτά τα ξέρουμε λόγω του στόχου του 2025 γιατί είναι πρώτον πυλών. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε από τεχνική σκοπιάς απόλυτα σωστά. Ο στόχος του 2030 με χαμηλότερη δυνατότητα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει πιστευτός. Ε, μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα έχουμε τεχνολογία τότε, αλλά πρέπει να προσέξουμε κάποιες λεπτομέρειες και θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες λεπτομέρειες. Καταρφάς, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συνεπώς το διοξίδιο του άνθρακα ανά χιλιόμετρο διότι αλλιώς θα έχουμε μικρότερα και λιγότερο αποτελεσματικά οχήματα. Και αυτό θα πρέπει να αντανακλείται και στον ορισμό των οχημάτων χαμηλών εκπομπών, που αυτή τη στιγμή ε, εκφράζεται με διοξίδιο του άνθρακα ένα χιλιόμετρο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια υποδομάδα για οχήματα υψηλών ε, επιδόσεων. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να έχουμε μακρύτερα οχήματα. Και για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ξεκινήσουμε από τον πιο χαμηλό στόχο και να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Τώρα, ε, Όσον αφορά τους διαβιβαστές, τους vectors, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Ε, να δούμε και αν ε, τα ε, στοιχεία που γίνονται σε δοκιμές στους δρόμους διαφέρουν από αυτά που έχουμε ως ε, ε, θεωρία. Ε, διότι αν είναι αλήθεια αυτό, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το θεωρητικό επίπεδο. Και αν επικαιροποιείται αυτό, τουλάχιστον ετησίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τους χαμηλότερους στόχου, για παράδειγμα οικολογικά χαρακτηριστικά. Τώρα, δανεισμό και τραπεζικά ζητήματα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε την έγκαιρη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους περιτούς το έχει κάνει πάρα πολύ περίπλοκο το όλο ζήτημα. Εάν κάποιος πουλά ένα φορτηγό, ή μάλλον το θέσω αλλιώς, αν τα πας καλύτερα, θα πρέπει να μπορείς να το χρησιμοποιείς ανα πάσα στιγμή στη διαδικασία. Το να αποφασίσουμε σε μηδενισμό των τάσεων ε, ε, των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα το 2025 σημαίνει ένα πράγμα, ότι ο κόσμος θα ε, παραπλανά το σύστημα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία παίρνει επιδόματα για τα παιδιά που έχει. Όσο περισσότερα ε, παιδιά έχει, ε, παίρνει περισσότερα χρήματα. Επομένω, ο κόσμο το βράδυ ε, κάνει προγραμματισμό με τα ημερολόγια του για να δει πότε θα κάνει το επόμενο παιδί. Ε, φτιάχνουμε και πολλά φορτηγά στη Σουηδία, επομένω κάπω έτσι θα τα σκεφτόμαστε. Ε, να το έχουμε λοιπόν ω στόχο και αν τα καταφέρουμε προχωράμε παραπέρα στην πορεία και κάνουμε την αλλαγή. Τώρα, καύσιμα χαμηλών εκπομπών. Κάναμε μεγάλη συζήτηση. Ε, το να λέμε χρησιμοποιήστε για παράδειγμα πυρηνικά απόβλητα δεν σημαίνει ότι θα έχουμε λύση. Ε, βιοκαύσιμα, ε, σε κάποιε περιπτώσει θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Κάποιοι ασχολούνται με τα βιοκαύσιμα, αλλά εμεί έχουμε αποφασίσει τι είναι σωστό και τι είναι λάθο με την οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά ήταν χωρί νόημα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί έχουμε την οδηγία. Και πρέπει να τα καταφέρουμε, γιατί αν δεν έχουμε την κατάλληλη ισορροπία, ε, σίγουρα θα ε, ζημιωθούν Ευρωπαίοι παραγωγοί και δεν θα πολλούνται νέα φορτηγά. Θα επισκευάζουν τα παλιά του φορτηγά. Και ένας λόγος είναι κυρίως το περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Φιέλνερ. Ο κύριος Τζόφολη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Επιτέλους, μπορούμε να το πούμε, επιτέλους μετά από χρόνια συζητήσεων, αναβολών, και αφού εγκρίναμε, να επενθυμίσουμε όλοι, το Μάιο, με πολλές συζητήσεις και αντιστάσεις, ε, την νομοθεσία για την παρακολούθηση και τη διαβίβαση των στοιχείων για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και της ε, κατανάλωση καυσίμων των νέων φορτηγών οχημάτων, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να καθορίσουμε και τα όρια για τις εκπομπές αυτών των οχημάτων. Μην ξεχνάμε δε ότι αυτές οι εκπομπές αποτελούν σήμερα το 6% των συνολικών εκπομπών και προβλέπονται απουσία παρεμβάσεων αυξήσεις μέχρι και 10% για το 2030. Πρόκειται λοιπόν για μια θεμελιώδη πρόταση για το σεβασμό των συμφωνιών των Παρισίων και να μην ε, ξεχνάμε και για να εξασφαλίσουμε σε πάνω από μισό εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων. Εξοικονόμηση καυσίμων που σημαίνει ότι τα καύσιμα θα συμβάλλουν κατά ένα τέταρτο στο λειτουργικό κόστος. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν ε, ταχύτατα η πρόταση κανονισμού αυτή και επομένως είναι ευπρόσδεκτη η ταχεία διαδικασία για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ διότι συνειδητοποιούμε ότι η διαδικασία ε, κάποια στιγμή θα εξεταστεί το 2022, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 13, θα υπάρξει αναθεώρηση. Επομένως, ε, ελπίζουμε ε, ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικά είναι καλή πρόταση, ισορροπημένη, λογική, δίκαιη, βάσει και της υπόδειξης δύο βημάτων. Το πρώτο το 2025 που είναι δεσμευτικός και το 2030 το οποίο θα υπόκειται σε παλήθευση. Εμείς ε, παρόλα αυτά θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ε, ώστε αν είναι δυνατόν η πρόταση να γίνει πιο φιλόδοξη. Και όσον αφορά τους στόχους, 20% για το 2025 και 35% για το 2030, τροπολογίες για να διευκρινιστεί ο ορισμός ε, του επαγγελματικού οχήματος, ο ρόλος των αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων και εδώ θα σταθούμε και ε, στην καλύτερη διευκρίνηση για την ενίσχυση των στόχων της επαλήθευσης και της αναθεώρησης το 2022, που είναι ουσιαστική στην όλη διαδικασία και βάση και ε, των κινήτρων που προβλέπεται με το σύστημα των σούπερ πιστώσεων. Αλλά για μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ο κανονισμός καταρχάς, ε, να ε, αναβάλουμε και πάλι αποφάσεις ε, ε, σημαίνει ότι θα καθυστερήσουμε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τις απαραίτητες συγκλήσεις, τις απαραίτητες ευελιξίες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επαναλαμβάνω, είναι ισορροπημένη. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε ώστε να έχουμε τον ηγετικό ρόλο σε βιομηχανικό επίπεδο στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα, την Ιαπωνία και τις Πολιτείες που έχουν ήδη καθορίσει όρια εκπομπών και το να υποστηρίξουμε, όπως λέγαμε, την έρευνα και την ε, ανάπτυξη στον τομέα θα δημιουργήσει νέες και καλές θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριος Μάθιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η ύβρις είναι το θανάσιμο αμάρτημα των πολιτικών. Κατεβαίνουμε σε εκλογές, υπερψηφίζουμε ψηφίσματα και περιμένουμε ο κόσμος να αλλάξει. Όμως ο πραγματικός κόσμος δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εμείς μπορεί να είμαστε εδώ και να συζητούμε για στόχους 15, 30, 45%. Μπορούμε να υπερψηφίσουμε και ψηφίσματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα συμβούν. Αυτά θα συμβούν μόνο αν υπάρχει η σχετική τεχνολογία και εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Όλα αυτά θα συμβούν αν ο στόχο είναι εφικτό, διότι αν είναι ανέφικτος δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Ό,τι και αν κάνουμε, όσο καλές ομιλίες και αν εκφωνούμε εδώ μέσα, στον πραγματικό κόσμο δεν πρόκειται να συμβούν όλα αυτά που λέμε. Συμφωνώ με τον Σουηδό συνάδελφο, με τα όσα είπε επί του θέματο, δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά είναι επίση σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι προσπαθούμε να προσδιορίσουμε του τρόπου με τον οποίο ο κλάδο ή οι πολίτε μπορούν να επιτύχουν του στόχους. Αυτό όμως είναι όμως επίσης μια ε, δύσκολη διαδικασία και δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι απλά. Πολύ συχνά πολιτικοί έχουν επιλέξει συγκεκριμένε τεχνολογίες που προωθούσαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες απεδείχθησαν αναποτελεσματικές. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα είναι ο κόσμος το 2050 ούτε, ούτε μπορούμε ακριβώς με τόση μεγάλη λεπτομέρεια να προβλέψουμε ή να θέσουμε στόχους διότι η τεχνολογία και ο κλαδο μπορεί να τρέξουν με διαφορετικούς Φυσικά υπάρχουν στόχοι ε, που ενδέχομένως ε, και να μπορούν να επιτευχθούν, αλλά ταυτόχρονα οι κατασκευαστές να επιλέξουν απλώς να πληρώσουν τα, τα πρόστιμα και αν υπάρξουν εμπορικά ωφέλη για τους ε, ανταγωνιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς τελικά δεν θα έχει κανένα όφελος, διότι το περιβαλλοντικό όφελος που θέλουμε να επιτευχθεί δεν θα έχει επιτευχθεί ούτε αυτό. Η ομάδα ECR θέλει να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε με τον κλάδο αλλά και με τους καταναλωτές προκειμένου να επιτευχθεί ότι είναι εφικτό και όχι να θέτουμε στόχους οι οποίοι είναι, ακούγονται ωραίοι και όμορφοι που μπορούν να κάνουν πρωτοσέλιδα, που μπορούν να πάρουν ακόμη και βραβεία αλλά που δεν πρόκειται να βοηθήσουν κανέναν και σε τίποτα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν πολύ στενά και πολύ προσεκτικά πώς θα προχωρήσει αυτή η πρόταση μέσα από το σύστημα. Ε, συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου ιδανικό. Το ζήτημα αυτό χρειάζεται προσεκτική εξέταση και μελέτη. Δεν μπορούμε να το διατρέξουμε έτσι στα γρήγορα λόγω ενός πολύ σφιχτού χρονοδιαγράμματος. Θέλουμε να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα. Θέλουμε να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι, αλλά θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ω προ τον τρόπο που θα επιτευχθούν αυτό. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να φύγω. Δεν θέλω ε, να με παρεξηγήσετε, αλλά δυστυχώς πρέπει να παρευρεθώ σε μια άλλη συνέδριση, συνέδριση η οποία έχει ξεκινήσει πριν από μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έκχουρτ και έχουμε ένα πλαίσιο εδώ το οποίο είναι φιλόδοξο και είναι οι δύο, η πρώτη προσπάθεια για, να, ε, για κάποια εναρμόνιση και για να υπάρχει κυκλοφορία χαμηλών εκπομπών. Ε, θα έχουμε βεβαίως και ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα επόμενα χρόνια από μεγάλους ε, αυτοκινητοβιομήχανους. Ε, πρέπει να... Βεβαίως δεν μπορούμε συνέχεια να μιλούμε για πάντα για μείωση μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Το μεσοπρόθεσμο είναι ήδη εδώ και πρέπει να ασχοληθούμε. Τούτων λεχθέντων έχουμε ευθύνη να, ε, να διορθώσουμε τα πράγματα και δεν πρέπει να έχουμε να εξαιρέσει νομίζω ότι τα πρότυπα ε, για επιδόσεων εκπομπών είναι σημαντικά ε, και θα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας σε σχέση με την πρόταση ε, της ε, Κομισιόν. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορες ε, προτάσεις και θα πρέπει να περάσουμε σε χαμηλότερα επίπεδα. Σκιώδης εισηγητής επίσης θα κάνει προτάσεις ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται με τις υποδομές. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ζητήσω από την Κομισιό για την Baseline 2019 και ε, μήπως αυτή η γραμμή έχει διονγκωθεί τεχνίτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκχάουτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Οι ακραίες καιρικέ συνθήκες που ε, ζήσαμε φέτος αποτελούν προάγγελους μιας περιβαλλοντικής και κλιματολογικής καταστροφής. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός ακόμη και αν υπάρχουν άνθρωποι που την αρνούνται ένθεν κακήθεν του Ατλαντικού. Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ήδη εδώ, γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε να αναλάβουμε δράση το συντομότερο δυνατό. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται ότι ξέχασαν τελείως τις κλιματολογικές επιπτώσεις των προϊόντων τους. Ξέχασαν και αγνόησαν τις ε, μοιραίες επιπτώσεις που έχουν στη ζωή μας και την υγεία μας τα προϊόντα τους. Οι νεκροί του περιβάλλοντος, των περιβαλλοντικών αλλαγών είναι, είναι περισσότεροι και θα είναι περισσότεροι από όσοι όλοι οι νεκροί όλων των, πολίτο, ε, όλων των πολέμων στην ιστορία του ανθρώπου. Μπορεί κανείς όλα αυτά να τα αγνοεί διότι για τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι σημαντικότερα τα κέρδη και τα μερίσματα των μετόχων από το να επενδύσουν τα χρήματα και τα κεφάλαιά τους στην καινοτομία και την έρευνα. Και δυστυχώς το φίδι γύρισε και δάγκωσε τις ίδιες αυτές αυτοκινητοβιομηχανίες διότι φαίνεται πλέον ότι η Κίνα και η Ιαπωνία πλέον είναι μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αυτοκινητοβιομηχανίες επέμεναν να λένε ψέματα στον κόσμο και ψέματα στον εαυτό τους. Εμείς σήμερα χρειαζόμαστε βιώσιμες συνθήκες για να εξασφαλίσουμε ε, ένα βιώσιμο περιβάλλον και για τις επόμενες γενιές. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε να καταλήξουμε σε περιβαλλοντική καταστροφή περιβαλλοντική καταστροφή τα επόμενα χρόνια. Συμφωνήσαμε στην, ε, στους στόχους των Παρισίων. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν έχουν ακόμη ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι αυτοί. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να ληφθούν δραστικά μέτρα για τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα τόσο στη γεωργία όσο και στις μεταφορές όσο και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μια μείωση των εκπομπών από τα φορτηγά κατά 15 ή 20% έως το 2015 ή 30% έως το 2030 είναι στόχος απαραίτητος ακόμη και αν συνοδεύεται από δυσκολίες όπως για παράδειγμα την γενική ε, κατασκευή σταθμών φόρτισης. Χρειάζεται όμως να γίνει γιατί κάτι τέτοιο θα επιφέρει και δημιουργία θέσεων ε, απασχόλησης. Βεβαίως λιγότερες σε αριθμό διότι η ηλεκτροκίνηση χρειάζεται ε, λιγότερους εργαζόμενους από την πετρελαιοκίνηση. Παρ' όλα αυτά, η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει επιτέλους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της και στο μέτρο που της αναλογεί στην κλιματική αλλαγή και να θέσει αυτό ως προτεραιότητα έναντι των κερδών της. Και η έκθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικότατο μήνυμα προς την αυτοκινητοβιομηχανία. βιομηχανία. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή που έχουμε. Εμείς ως πολιτική ομάδα και εγώ προσωπικά πάντως βρισκόμαστε απολύτως στο πλευρό του εισηγητή και σας συγχαίρω για το κείμενό σας. Ωραία. Η κυρία Εύνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ παίρνω το λόγο για το θέμα αυτό. Χαίρομαι που μπορούμε επιτέλους να το συζητήσουμε με τους αδέλφους. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει να καθορίσει πρότυπα για τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων, ελπίζοντας να μειώσει το χάσμα που υπάρχει με άλλες περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία ή και η Κίνα, ε, στις οποίες έχουν ήδη εγκριθεί μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε και σε μια ευνοϊκή περίοδο διότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε επικοδομητικά για τον κανονισμό, για την ε, ε, πιστοποίηση και να έχουμε και καλά αποτελέσματα σαν αυτά τα οποία καταφέραμε στον κανονισμό για την παρακολούθηση και τη διαβίβαση των στοιχείων που αφορούν ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων που εγκρίναμε πρόσφατα τον Ιούνιο, πάντα για τα βαρέα οχήματα. Διότι ε, το γεγονό ότι οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα των λεωφορείων και των φορτηγών μέχρι τώρα δεν έχουν ρυθμιστεί, οδήγησε ε, σε προβλήματα και έχουμε προβλήματα ω συνομοθέτε, τα οποία θα πρέπει να προλάβουμε ε, και να υπάρχει ε, πρόληψη γενικότερα. Χωρίς μέτρα, το είπαν οι συνάδελφοι, οι εκπομπές θα αυξηθούν κατά 9% το διάστημα 2010-2030 λόγω της αύξησης των ε, μεταφορών. Και επίσης, αυτό θα ήθελα να το τονίσω, η αρμόδιοι στον τομέα των μεταφορών δεν θα μπορέσουν να έχουν κανένα πλεονέκτημα στην οικονομία κλίμακα όσον αφορά την κατανάλωση και το κόστο του καυσίμου, που θα μπορούσε να προκύψει αν έχουμε κάποια πρότυπα μείωση σε αυτή την περίπτωση. Κατά την άποψή μου, είναι απαραίτητο να επιλέξουμε επίπεδα μείωση εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα που θα εγγυώνται τις μεγαλύτερες καθαρές απολαβές ε, και ε, οικονομίες ε, μέχρι το 2030 και ε, να μπορέσουμε να έχουμε μία αποφασιστική στροφή προς την ηλεκτροκίνηση και για αυτά τα οχήματα. Διότι σήμερα η παρούσα κατάσταση, άκουσα τις διάφορες απόψεις των συναδέλφων, κατά την άποψή μου είναι παράλογη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ε, τεχνολογίες αυτή τη στιγμή σήμερα, οι οποίες χρησιμοποιούνται και μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του καυσίμου κατά 18% οδηγώντας σε εξοικονόμηση του απίστευτου ποσού των 5.700 ευρώ το χρόνο. Και ε, δεν υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή δεσμευτικά πρότυπα και είναι και αποτυχία της αγοράς που δεν επιτρέπουν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι αυτά προτείνονται ο μόνος προαιρετικά μέτρα και αυξάνεται δυσανάλογα και το κόστος αγοράς αυτών των οχημάτων. Κατά την άποψή μας αυτό δεν είναι πλέον αποδεκτό και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθορίζοντας ε, κάποιους στόχους ε, φιλόδοξης μείωσης όπως ε, ζητήσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ζήτησαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ε, logistics και μεταφορέων που προτείνουν μείωση κατά 24% για το 2025 και ε, δεσμευτικές ε, μειώσεις στα φορτηγά μηδενικών εκπομπών. Κατά την άποψή μου, η μείωση ε, των τιμών των βαρέων οχημάτων με χαμηλέ και μηδενικέ εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να μειωθεί κατά 25% και θα πρέπει και το 2025 να έχουμε φτάσει ε, σε περικοπή ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στο 20% τουλάχιστον μέχρι το 2025. Πρέπει να δεχτούμε την ηλεκτροκίνηση ω επιλογή και για τον τομέα των βαρέων οχημάτων, όχι μόνο γιατί το ζητούν οι αρμόδιοι του κλάδου, αλλά και γιατί είναι ακόμα σαφή η επιλογή πολλών ε, ευρωπαϊκών πόλων οι οποίες προσπαθούν να ε, μην έχουν τεχνολογία δίζελ και οχήματα δίζελ τα οποία να κυκλοφορούν στους δρόμους τους διότι αυτό οδηγεί στα γνωστά προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης τα οποία δεν είναι αμελητία σε καμία περίπτωση. Η πρόταση της έκθεσης του συναδέλφου Χάουτ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Εκτιμούμε και τις προτάσεις του εισηγητή, ο οποίος ζητά να αυξηθεί ουσιαστικά η μείωση των στόχων και για το ε, διάστημα μέχρι το 2029 και για το διάστημα μετά το 2030 και εγώ ως και εισηγήτρια θεωρώ ότι για να ε, εξασφαλίσουμε τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές θα πρέπει να καθορίσουμε ε, στόχους ε, ελάχιστης ε, παραγωγής για το στόλο κάθε παραγωγού και για το 2025 και για το 2030, προσφέροντας ευελιξία στους κατασκευαστές οι οποίοι θα μπορούν να αποφασίσουν τι επενδύσεις θα κάνονται, πριμοδοτώντας βεβαίως αυτούς οι οποίοι θα δράσουν πρώτοι. Θα υποβάλουμε και εμείς τροπολογίες και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε λοιπόν με τους σκιώδεις εισηγητές, κυρία Αγιούς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να τον συγχαρώ για τη δουλειά του. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ισορροπημένη και ρεαλιστική κατά την άποψή μου Βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Σάικχαουτ, το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο. Είναι αλήθεια ότι από τεχνική σκοπιάς ε, υπάρχει δυνατότητα στο εγγύς μέλλον ε, να καταφέρουμε κάποια πράγματα, αλλά όπως είπε και ο κύριος Φιέρνερ, αυτό θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Και επομένως θα οδηγήσει σε αγορά λιγότερων οχημάτων το κόστος ε, κατασκευής, που είναι το πρόβλημα, θα ε, μεταβιβαστεί ε, στον καταναλωτή. Αυτό γίνεται πάντα. Επομένω πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι μεν, αλλά να τα σκεφτούμε κιόλα. Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά τις προτάσεις ευελιξίας και την εφαρμογή της τεχνολογικής ιδιωτερότητας. Τα πάντα έχουν σημασία εδώ και όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι εξαιρετικά γιατί δεν έχουν εκπομπές. Αλλά ένα ηλεκτρικό όχημα είναι μπαταρία με ρόδε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όλο το πλαίσιο. Πρέπει να κατασκευαστεί μπαταρία. Εκπέμπονται πολλά για την κατασκευή μιας μπαταρίας, πάρα πολλά. Οι μπαταρίες αυτές έχουν και περίοδο ε, στην οποία δεν λειτουργούν ε, όπως ε, γίνεται και με τα τηλέφωνα. Στην αρχή λειτουργούν καλύτερα και σιγά σιγά η μπαταρία ευθύνει. Επιμένως πρέπει να σκεφτούμε και το τέλος ζωής των μπαταριών, ανακύκλωση κλπ. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε όλο το πλαίσιο διότι αλλιώς εφαρμόζουμε το νόμο του εκκρεμούς. Και μπορεί να γίνει ό,τι έγινε με το ντίζελ και, το, και τη βενζίνη. Ε, προσπαθούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, επιλέγουμε τον ντίζελ και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε εκπομπές ε, υδρογόνου και θέλουμε να εγκαταλείψουμε τον ντίζελ. Επομένως θα ήθελα να ζητήσω να αναλυθούν τα πάντα και να το ζητήσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και να είμαστε ρεαλιστές ε, και η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ κυρία Γιούσο. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει τον λόγο πάνω στο θέμα αυτό. Εάν όχι, τότε δίνω τον λόγο στην Επίτροπη. Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Κομισιό και ευχαριστώ επίσης τον εισηγητή για την πρόταση και για όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Το πρώτο πράγμα που συγκρατώ είναι ότι ε, οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, διότι ξέρουμε ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, οι εκπομπές αυτές θα αυξηθούν. Θέλουμε να βεβαιωθούμε και αναφέρθηκαν κυρίως οι καταναλωτές, οι χρήστες, ε, να κατανοήσουν ε, την ε, σημασία εξοικονόμησης εκπομπών με τα βαρέα οχήματα επαγγελματικά και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ε, να μείνουν στο προσκήνιο διότι αυτοί είναι οι καινοτόμοι και θέλουμε το εμπόδιο να το βάλουμε λίγο ψηλότερα για αυτούς ούτως ώστε να είναι καλύτερος ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός που απειλείται. Εξετάζοντας την πρόταση της Κομισιόν βλέπουμε ότι είναι ε, την πρώτη ε, φορά που ασχολούμεθα με τις εκπομπές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και θέλουμε όλοι ε, να έχουν μια ε, εξέταση για να έχουμε αναθεώρηση το 2022. Δεν έχουμε ακόμα την baseline, τη βασική γραμμή ε, και που θα έρθει με την πρόταση που υιοθετήθηκε πρόσφατα για το monitoring, την παρακολούθηση και θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε και αυτό έχει σχέση με το θέμα που αναφέρθηκε από τον κύριο Τόρμπας ε, λέγοντας ότι μπορούν οι κατασκευαστές ε, να ε, ασχοληθούν με τις, τα στοιχεία 2019. Βεβαίως οι ευφύς μηχανικοί μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά και ο κύριος Φέρνα αναφέρθηκε ώστε ότι πρέπει να εξετάσουμε το Vector. Το Vector είναι ένα νέο εργαλείο το οποίο θα δοκιμαστεί πραγματικά τα επόμενα χρόνια και πρέπει να δούμε ποιος θα αποδώσει και θα πρέπει να ενημερωθεί, να επικαιροποιηθεί, διότι νέες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν και ε, οικονομικά μόνο θα μπορέσουν να καλυφθούν ορισμένες σειρές βαρέων οχημάτων. Ε, τα οχήματα αυτά καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, ε, γι' αυτό είναι σημαντικές οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και είναι σημαντική επίσης η εξοικονόμηση καυσίμων. Οι στόχοι που προτάθηκαν η Κομισιό βάσει της αξιολόγησης αντικτύπου ε, διάβασα πολλές φορές πρόκειται για στόχους φιλόδοξους και για να εξηγήσω το 15 ως 20% βέβαια το 20% θα επιτευχθεί ε, όταν όλα λειτουργήσουν καλά ταυτόχρονα και όσο προς τις υφιστάμενες τεχνολογίες αν τις εξετάστε, υπάρχουν μερικοί κατασκευαστές που έχουν ορισμένες άλλοι έχουν άλλες ενώ υπάρχουν στη διάθεση όλων. Νομίζουμε ότι 15% είναι φιλόδοξο στόχος, ο κύριος Μάθιους δεν είναι πλέον εδώ. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι φυκτό, επιτεύξιμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ασχοληθήκαμε στην πρόταση με ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, ενώ ε, ε, υπάρχει ε, πρόταση να περάσουμε σε άλλες σειρές. Ίσως λόγω έλλειψης στοιχείων ήταν αδύνατον για μας να κάνουμε μελέτη αντικτύπου, αλλά θέλουμε να επανέλθουμε στις κατηγορίες αυτές οχημάτων το 2022, ε, τις, τις μικρές καμιονέτες, ε, τα πούλμαν, τα λεωφορεία, για να δούμε τι είδους τεχνολογίες έχουμε, θα έχουμε διαθέσιμες ε, τα επόμενα έτη. Μερικοί παρατήρησαν ότι για τα λεωφορεία. Η τεχνολογία προοδεύει αρκετά ε, γρήγορα και θα πρέπει ε, στην αξιολόγηση αντικτύπου 2022 να το δούμε αυτό. Έχουμε λοιπόν κίνητρα ε, για τα οχήματα με χαμηλές εκπομπές και μηδενικές εκπομπές. Μπορούμε βεβαίως να αναθεωρήσουμε την κατάσταση το 2022 αν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, αλλά αν θυμηθείτε όταν εισήχθη η νομοθεσία για τα ε, αυτοκίνητα αρχίσαμε με τα super credits και περάσαμε ε, σε αυτές τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά το, την, ε, το λόγο κόστους ωφέλους υπάρχει κάποια ευελιξία λόγω της ειδικής ε, δομής ε, των ε, φορτηγών που είναι διαφορετικά από τα αυτοκίνητα. Ήταν σημαντικό να σκεφτούμε τις τράπεζες, τον δανεισμό και ως προς την διακυβέρνηση κάναμε, εξετάσαμε παράλληλα και νομίζουμε ότι μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι κατασκευαστές θα επιλέξουν νέες τεχνολογίες και όχι απλώς θα πληρώσουν το πριμ που όπως μερικοί είπαν και αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση ότι είναι ψηλό το επίπεδο αυτό που βρίσκεται στην πρόταση. Σχετικά με τις υποκείμενες τεχνολογίες Έχουμε μελετήσει τι έχει γίνει για να εξετάσουμε τις διάφορες τεχνολογίες και θα δημοσιευθούν αυτές οι μελέτες στις επόμενες δύο εβδομάδες. Προ, ε, σύντομα, δηλαδή προσεχώς, δεν ξέρω ακριβώς αν θα είναι σε δύο εβδομάδες, για να δούμε ε, τι υποθέσεις έχουμε λάβει υπόψη για την μελέτη αντικτύπου. Νομίζω ότι είναι μια ενδελεχής μελέτη που προσπαθεί να είναι πάρα πολύ ρεαλιστική εξετάζοντας τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Εξετάζοντας ένα τελευταίο θέμα που είναι το θέμα των καυσίμων, νομίζω ότι από πλευράς της Κομισιό ίσως αντίθετα με την κατάσταση με τα αυτοκίνητα πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα όταν πρόκειται για τα φορτηγά, ε, τα, τα φορτηγάκια ε, τα, και που έχουν, καλύπτουν μικρές αποστάσεις κάθε μέρα, αλλά όταν πρόκειται για τις μεγάλες αποστάσεις, τα οχήματα που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, θα πρέπει να δούμε τα βιοκαύσιμα και αν θα μπορούμε να έχουμε απανθρακοποίηση και έχουμε κίνητρα ε, με την οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα που αποφασίστηκε από τους συνομοθέτες και νομίζω ότι εξετάσαμε αν θα έπρεπε αυτό να περιληφθεί ε, στα ωφέλη ε, που περιλαμβάνονται στην πρόταση και έχουμε καταλήξει στην ίδιο συμπέρασμα με τα αυτοκίνητα ότι δεν πρέπει να υπάρχει διπλή καταμέτρηση это ε, η ευθύνη ανήκει στον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν ξέρουν ε, τι ο οδηγός του φορτηγού ε, χρησιμοποιεί, αν είναι βιοδίζελ, βιοαέριο και από αυτήν την άποψη ακολουθούμε τον ίδιο ε, τρόπο ε, που ακολουθήσαμε στην πρόταση για τα αυτοκίνητα. Μακρηγόρησα ίσως, αλλά ελπίζω ότι ήταν χρήσιμα τα όσα σας είπα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έικχαουτ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης και τους άλλους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι με βοηθούν πολύ, καθώς και την ε, Κομισιόν για τις εξηγήσεις που μας έδωσε αλλά και την υπόσχεση να μας παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Και αυτό είναι σημαντικό διότι αν κατάλαβα καλά τον Κρίστοφερ αν στα λιπαντικά μπορούν να συμβαίνουν αυτά ε, τότε θα αλλάξει και η καριέρα από ό,τι μας είπε. Αυτό καλό θα είναι. Ναι, ναι, και θα πλουτίσεις βεβαίως. Να, σημειωθεί και στα πρακτικά βεβαίως ότι, ότι αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, συνοψίζοντας, να πω τα εξής. Η συζήτηση θα... Ε, μας απασχ... Στην συζήτηση θα μας απασχολήσουν τα εξή. Βεβαίως, ο εξηλεκτρισμός είναι ένα ζήτημα, είναι μια νέα τεχνολογία που θα πρέπει να λάβει και ε, κίνητρα ε, και υπάρχει, υπάρχουν ακόμη και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο τεχνολογιών. Όσον αφορά το 15-20% μείωση, βεβαίω ο στόχο αυτό αφορά και τη βελτίωση τη υπάρχουσα τεχνολογία, αλλά και την ανάγκη προετοιμασία, ώστε μετά το 2025 πραγματικά να, να προχωρήσουμε σε μια απότομη μείωση των εκπομπών. Και αυτό είναι ο βασικό μα στόχο. Βεβαίω, άκουσα και κάποιον συνάδελφο να λέει ότι θα ήθελε υψηλότατα ε, super credits, ο Νίλης νομίζω ε, είπε ότι έχει κάποιες ε, αμφιβολίες σε σχέση με αυτά τα super credits, αυτές τις υπερπιστώσεις. Είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η εντολή που δίνουμε είναι μετριοπαθής και αυτός είναι και ο καταλληλότερος τρόπος. Γιατί υπάρχουν και χωρία στη μελέτη αντικτύπου οι οποίες μας, τα οποία μας επιβεβαιώνουν ότι ορθώς ακολουθούμε αυτήν την πορεία. Βεβαίως υπάρχουν και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Να υπενθυμίσω όμως ότι η εντολή μας αφορά χαμηλές και μηδενικές εκπομπές. Ποιος είπε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Κανείς δεν το είπε αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι ως προς το διεξίδιο του άνθρακα, και θέλουμε ταυτόχρονα να πούμε ότι ε, χρειαζόμαστε και μικροπιστώσεις, ε, σούπερ πιστώσεις, συγγνώμη, τότε ε, στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Χρειάζεται, αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε και να καταργήσουμε τις εκπομπές, πρέπει να ε, παλέψουμε σε όλα τα μέτωπα. Καλέ είναι οι προτάσει που έχουν γίνει, αλλά αν συμφωνούμε πραγματικά όλοι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν και στην πράξη, και μάλιστα το επιβεβαίωσε αυτό και ο συγητή του ΕΛΚ, ε, τότε α μην διαμαρτυρόμαστε ότι προσπαθούμε πραγματικά να αναλάβουμε δράση σε διάφορα μέτωπα. Όσον αφορά την γραμμή αναφορά για το 2019. Αυτή ακριβώς είναι και η βάση που χρησιμοποίησαμε για τις αλλαγές που προτείναμε. Προσπαθήσαμε δηλαδή να ε, μετριάσουμε αυτόν τον, αυτούς τους κινδύνους και επίσης κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του βραχυπρόθεσμου και του μακροπρόθεσμου ε, επίπεδου. Διότι όπως υπόθηκε και νωρίτερα, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι το 2025, βεβαίως μπορούμε να δείξουμε κάποια ευελιξία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχεις ξεπεράσει τους στόχους που, που έχεις θέσει για το 2030. Τέλος. Θέλουμε αυτή η διαδικασία να ενταχθεί και στην διαναθόρηση του 2022. Βεβαίως. Και αυτό το θέμα ε, πρέπει να, πρέ, οι διαδικασίε μα και οι στόχοι μα πρέπει να αναθεωρηθούν το 2022, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2022, ιδίω για τα λεωφορεία. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε η νέα Κομισιόν να διεξαγάγει μια νέα μελέτη αντικτύπου και να φτάσουμε μέχρι το 2022 για να δούμε τι έχει γίνει. Πρόκειται για σπατάλη χρόνου. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι σπατάλη χρόνου. Πρέπει από τώρα να λάβουμε δράση ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Και βεβαίως στη συνέχεια να, γίνουν και, να γίνει και ένα θεώρηση το 2022 η οποία όμως θα έρθει να δει αν τα πράγματα δεν πήγαν καλά όχι να περιμένουμε να αναλυθεί η δράση το 2022, διότι αυτό, όπως είπα, θα είναι σπατάλη χρόνου. Και να υπενθυμίσω και αυτό που είπε ο κύριο Εκ, ότι δεν έχουμε τον, την πολυτέλεια του χρόνου ούτε από άποψη κλίματο ούτε από άποψη καινοτομία. Διότι άλλε περιφέρειες, άλλε χώρε στον κόσμο έχουν ήδη τέτοιου στόχου για τα βαρέα οχήματα. Είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε ουραγοί σε αυτό το τομέα. Δεν θα χάσουμε λοιπόν μόνο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά θα χάσουμε και στον τομέα τη καινοτομία. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το χειρότερο που μπορεί να μα συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Προθεσμία, όπως είπε και ο κύριος Φιέλνερ, είναι πολύ σύντομη. 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε όμως ε, ε, εξοικείωση με τη συζήτηση των ίδιων θεμάτων. Ίσως λοιπόν να έχουμε χρόνο. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν προθεσμία για τις κατα... τροπολογίες. 18 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην ΕΜΒΗ. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης, που είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπταξης και το Ταμείο Συνοχής. Εδώ εξετάζουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Συντάκτρια είναι η κυρία Κονέτσνα. Έχετε το λόγο. Děkuji, paní předsedkyně, ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο λόγια για τη γνωμοδότηση. Όπως γνωρίζετε, στις 2 Μαΐου εγκρίθηκε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση 2020-2027 που περιλαμβάνει και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απλοποιεί κάποιες διαδικασίες και για το Ταμείο Περιφερειακής Ενάπταξης και για το Ταμείο Συνοχής και διευκρινίζει και κάποιες διατάξεις για κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Ε, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι επενδύουν περισσότερο σε μια Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άρθρακα, ε, κυρίως όσον αφορά την κυκλική οικονομία, την ε, ε κυκλοφορία έξυπνων συστημάτων ενέργειας, ε, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ε, μείωση της ρήπανσης και βελτίωση της βιώσιμης χρήσης των υδάτων κλπ. Αυτά ανταποκρίνονται στις ε, σημαντικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και επομένως ε, θεώρησα ότι πρέπει απλώς να θίξω κάποια σημεία που είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ελπίζω. Πρέπει καταρχάς να έχουμε περισσότερους φόρους για τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους νέους φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον, τις μεταφορές, ε, τα απόβλητα και το κλίμα, σεβόμενοι και τις δεσμεύσεις του Συμφωνίας των Παρισίων. Ε, μεταξύ άλλων βεβαίω δημιουργούνται και πολλές θετικέ εργασίες στι διάφορες περιφέρειες και μειώνει τι κοινωνικές ανισότητες. Η χρήση αυτών των δύο ταμείων είναι το 50% των δημοσίων επενδύσεων. Χωρί λοιπόν αυτού του πόρου Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ε, χρηματοδοτήσουν αυτέ τι επενδύσει. Ε, τα κονδύλια του Ταμείου συνοχή θα χρησιμοποιηθούν για ε, προγράμματα για το περιβάλλον και το κλίμα, για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μείωση των ταμείων αυτών στην ε, διαχείριση δεν είναι σωστή. Θα πρέπει να συνδέσουμε τις επενδύσεις με τα σχέδια των κρατών μελών όσον αφορά το σεβασμό των στόχων για το 2030 και αυτό αφορά και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 5% ε, σε πόρους για τον ε, στρατηγικό στόχο 2 και επειδή πρέπει να μειώσουμε ουσιαστικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δεν μπορούμε να έχουμε καθυστερήσεις. Προτείνω λοιπόν να προωθήσουμε την αστική κινητικότητα ε, με συνδυασμένες μεταφορές που αυτή τη στιγμή στο στόχο 3 που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περάσει στο στόχο 2. Υπάρχουν περισσότεροι πόροι και αποτελεί ε, μεγαλύτερη πίεση λοιπόν ε, για τα κρατημένα παραμείνει εκεί. Ε, δεν υπάρχουν υποδομές ε, για την αστική κινητικότητα. Η πλειοψηφία των ε, σταθμών ανεφοδιασμού ε, βρίσκεται μόνο σε τρία κράτη-μέλη που αποτελούν το 37% ε, των κρατών μελών. Επομένως, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών και ε, χάρη σε κοινοτικούς πόρους. Φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε και μεγάλες περιόδους ε, ξηρασίας, ε, πυρκαγιές ε, και πλημμύρες. Και μάλιστα οι πλημμύρες σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο φέτος. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τι γίνεται με τους υδάτινους σπόρους εν γέννη. και να εξυγχρονίσουμε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πλέον απαρχαιωμένες και δεν μπορούν να βοηθήσουν για την επεξεργασία των υδάτων και την επεξεργασία των ε, λιμάτων. Πρέπει λοιπόν ε, να βοηθήσουμε να προχωρήσει και η κυκλική οικονομία, να διευκολύνουμε την πρόσβαση ε, στον τομέα της υγιεινής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συζητήσεις για τα διάφορα σημεία και περιμένω σχόλια όχι μόνο από τους κοιόδης συντάκτες, αλλά από όλους. Είμαι ανοιχτή σε διάφορες παρατηρήσεις και θα ακούσω ό,τι παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τουρκάνου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τολμηρή αυτή απόπειρα να πλουστεύσει τη διαδικασία και γιατί ε, έθεσε υπό την ίδια σκέπη διάφορα προγράμματα όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα δύο ταμεία που συζητάμε σήμερα. Το, το Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη και το Ταμείο Συνοχή είναι δύο προγράμματα χρηματοδότηση, τα οποία είναι ε, συνολικά και ε, σύνθετα και υπάρχει και ε, πολύ σημαντική χρηματοδότηση στο πλε... παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαι απογοητευμένο που η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνει τα κονδύλια τα οποία θα πάνε στα δύο ταμεία κατά το ίμιση και συμφωνώ με την κυρία Κονέτσνα ε, η οποία προτείνει ότι οι μειώσεις ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλες. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση κονδυλίων θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως περικοπές στη χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ε, πορεία των ε, προγραμμάτων και καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη θεματική συγκέντρωση για τους πέντε πολιτικούς στόχους, μετάβαση σε μη ρηπογόνες, επενδύσεις, ανάπτυξη, κινητικότητα και διασύνδεση των περιφερειακών μεταφορών σημαίνει προώθηση ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, και ε, διασυνδεδεμένη ανάπτυξη αστικών περιοχών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική στόχη. Και όσον αφορά την ανάπτυξη των περιφοριών υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η καταπολέμηση των περιφερειακών διαφορών και ανισοτήτων θα πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αντιμετωπίζουν διάφορες ε, καταστάσεις και η γεωπολιτική κατάσταση μιας περιοχής έχει και αυτή τη σημασία της. Εννοώ δηλαδή ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούμε περισσότερο τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές ε, και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι οι ανατολικότερες περιοχές στα σύνορα με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να έχουμε για την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Θα πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν υποδομές και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει βαθμολόγηση όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Η συγκεκριμένη πρότασή μου λοιπόν είναι να δώσουμε προτεραιότητα σε επενδύσεις σε περιοχές ε, που το ΑΕΠ είναι χαμηλό, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να συναισθανθούν και αυτοί ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απτά ε, αποτελέσματα. Το 20% των περιοχών που ανέφερα χρειάζονται κατεπηγόντως επενδύσεις σαν αυτές που σας ανέφερα. Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι το 50% ε, των δημόσιων επενδύσεων και χρειάζονται διακαώς ε, τα κρατημέλη αυτές τις επενδύσεις για να μπορέσουν να αναπτύξουν και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας ε, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των περιφερειών. Η έκθεση της κυρίας Κονέντσνα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία αφορά τους σταθμούς ανεφοδιασμού για τα οχήματα χαμηλών εκπομπών, ε, τροπολογίες 1 και 2. Θα αποτελέσει προτεραιότητα και την ευκαιρία για τις ανεπτυγμένες περιοχές κάτι τέτοιο. Άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο σε άλλες μάλλον περιοχές που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες, δεν αποτελεί απορρετήτως προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια μέση οδό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και προσαρμογές ε, στις ανάγκες των ε, περιφερειών που συμμετέχουν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μας και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να διαχειριστούμε και ε, ε, περίοδους ξηρασίας. Η πολιτική συνοχή είναι ουσιαστική για την πραγματική κυκλική οικονομία και λιγότερο αναπτυγμένε χώρε θα πρέπει να έχουν και αυτέ τη δυνατότητα να βελτιώσουν την επεξεργασία των ε, αποβλήτων και τις σχετικές εγκαταστάσεις ή θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάσουν νέες τέτοιες εγκαταστάσεις ε, όπου δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών Δεδομένου ότι και τα νοσοκομεία στις λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχές δεν έχουν ε, λάβει επενδύσεις και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και κυρίως την πτυχή της υγείας και των ε, πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει ε, κατά την άποψή μου να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, επιτρέποντας ε, σε πρόσβαση σε ευέλικτη χρηματοδότηση, η οποία θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας εκ μέρους Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για το έργο της. Προφανώς δεν αμφιβάλλει κανείς για την αξία της πολιτικής συνοχής. Δυστυχώς ο προϋπολογισμός των ταμείων αυτών μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο. Πέραν όμως από την ενεργειακή αποδοτικότητα, την προσερμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, τη διατήρηση και τη διαχείριση της βιολογικής ποικιλότητα πρέπει να ε, προσθέσουμε στους στόχους αυτούς και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο τα βιώσιμα έργα, τα πράσινα έργα να λάβουν προτεραιότητα όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων. Υποστηρίζω την πράσινη χρηματοδότηση και πιστεύω ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε αυτήν την αρχή. Πιστεύω ότι οι επενδύσεις στην ιατρική έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από ό,τι έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Προσλέγω στην καλή συνεργασία και με την συγκίτρια και με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρίσπο αντικαστά την κυρία Ρικιμάκη. Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει χρήματα στους τομείς που υπόσχονται τα περισσότερα στην οικονομία και περισσότερη μείωση εκπομπών ανθρακούχων και σε αυτούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και για να υπάρξει ανεξαρτησία από τις επιδοτήσεις. Θα πρέπει να πλουστευτεί η γραφειοκρατία στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει των δύο ταμείων οι στόχοι να συμφωνούν με την συμφωνία του Παρισιού. Ε, νομίζω ότι η συγγήτρια ε, ασχολήθηκε πολύ καλά με την ε, υποδομή των μεταφορών και τις προκλήσεις. Υπάρχει ένα θέμα, θέλει η Συγήτρια να τοποθετήσει την πολυτρο, τις πολυτροπικές μεταφοράς μέσα στο πλαίσιο αυτό ή μόνος έναν τρόπο και θα πρέπει τότε να υπάρχει ένας στόχος που να καλύπτει όλες αυτές τις μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ που υποβλήθηκε αυτό το σχέδιο κειμένου σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με την εισηγήτρια και με την χρήση των πόρων που προτείνει που δεν λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα βεβαίως να ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή και πολύ συχνά αγνοεί το σχέδιο που προστατεύει το περιβάλλον και που ενθαρρύνει στην σπατάλη πόρων. Η ε, κυκλική οικονομία είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Επιτροπής μας σε αυτή τη θητεία και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε ό,τι περιλαμβάνεται στο πακέτο κυκλικές οικονομίας. Πώς θα γίνει αυτό στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Ταμείο Συνοχής. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν ε, τους στόχους που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και της ποιότητας ζωής των πολιτών τα ταμεία αυτά θα πρέπει να είναι κινητήρες αλλαγή να επιτρέπουν να προσανατολιστεί ο ιδιωτικό τομέας για να προσαρμόσει ε, το μοντέλο του. Έτσι θα έχουμε κοινού στόχου, αλλά είναι ε, κρίσιμο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί πόροι για να δούμε αν είμαστε στον καλό δρόμο. Εξ ονόματος της Κομισιόν τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που μου δίνεται να λάβω τον λόγο σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την επικοδομητική προσέγγιση και την αναγνώριση των προσπαθειών της Κομισιόν για την μεγιστοποίηση της πολιτικής συνοχής ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακος. Οι ε, δύο δηλαδή, ταμεία είναι στοιχεία κλειδιά σε αυτήν την συμβολή μιας τέτοιας ανάπτυξης και ενδεκτικά ποσοστά στα οποία εστιαζόμαστε ε, για μια πιο πράσινη Ευρώπη είναι πιο ψηλά από το μέσο όρο που παρουσιάστηκε ε, στον προϋπολογισμό ε, της Κομισιόν για μετά το 2020 λόγω των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν οι πόροι αυτοί και έχουμε τα παραδείγματα που μας δώσαν αξιότιμα μέλη σήμερα το απόγευμα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά σημεία, αν μου το επιτρέπετε, σχετικά με την οδομή των κανονισμών. Έχουμε έναν από τον κανονισμό για, για κοινή ε, και διαχείριση πόρων εκτός από τις ειδικούς κανονισμούς ε, για ε, τα σπόρους υπάρχει ο γενικός κανονισμός για τις γενικές διατάξεις που περιλαμβάνει πάρα πολλές λεπτομέρειες για την συντονισμό μεταξύ των ταμείων που αναφέρθηκε και επίσης έχουμε μερικά ε, στοιχεία για τα οποία εκφράστηκαν ανησυχίε σχετικά με τις προσπάθειες συγκέντρωση της χρηματοδότησης. Οι περισσότερες από αυτές τι λεπτομέρειες είναι στον κανονισμό γενικών διατάξεων και όχι στους κανονισμούς ξεχωριστά για το κάθε ταμείο. Γι' αυτό θα ήθελα ε, να μην υπάρχει ανησυχία θα έχουμε μετά το 2020 με βάση αυτή την πρόταση μεγαλύτερο μερίδιο για το Ταμείο Συνεχής. Θα υπάρξει αύξηση συγκέντρωσης για τις δαπάνες. Το τελευταίο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι θα δείτε ότι το κείμενο αυτού του κανονισμού είναι αρκετά σύντομο και αυτό ήταν μια επιλογή που κάναμε. Προσπαθούμε ως μέρος της απλούστευσης να μειώσουμε τα κείμενα, την νομοθεσία και μπορέσαμε να περικόψουμε τους κανονισμούς κατά το ίμιση όσον αφορά τον αριθμό των λέξεων. Βεβαίως αυτό δεν είναι απλούστευση αυτόματα, αλλά νομίζουμε ότι σε μεγάλο μέρος είναι και προσπαθούμε να αποφύγουμε να αναφέρουμε ε, υπερβολικές λεπτομέρειες ε, στις δραστηριότητες που μπορούν να υποστηριχθούν. Βεβαίως, ένα από τα σημεία για το Ταμείο Συνοχής είναι η κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη και της περιφέρειας. Δεν θέλουμε ε, να έχουμε υπερβολικές λεπτομέρειες στο επίπεδο του κανονισμού για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ευελιξία ούτως ώστε τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να μπορούν να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους με τον καταλληλότερο τρόπο ε, ακολουθώντας τις προτεραιότητες τους. Αυτό εξήγει καμιά φορά γιατί δεν έχετε όλα τα επίπεδα ε, λεπτομεριών. Έχουμε ορισμένα παραδείγματα ε, που εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την υποστήριξη στην υγεία, στην κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι παρούσα εδώ και η υγεία. Αυτό που δεν κάναμε όπως στο παρελθόν είναι να αναφέρουμε πάρα πολλά λεπτομερή παραδείγματα. Αυτή ήταν επιλογή μας για να έχουμε τον, ε, το πλαίσιο για την κατάλληλη ευελιξία όταν γίνεται η επιλογή των προγραμμάτων. Αυτό εξηγεί την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κονέτσινα. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη συζήτηση. Είμαι ανοιχτή σε διάφορες απόψεις και χάρηκα αυτή τη ε, ε, συζήτηση. Σίγουρα θα υπάρξει χρόνος να συζητήσουμε όλες τις διάφορες ε, μετακινήσεις κονδυλίων στις συνειδριάσεις των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. 5 ε, Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών και ψηφοφορία στις 18 Οκτωβρίου. Περνάμε στο τελευταίο σημείο. Εξέταση σχεδίου έκθεσης για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Γεωργίας αποφάσισε να επισπεύσει την ψηφοφορία της και έτσι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να ε, συντάξουμε μια γνωμοδότηση είναι να επισπεύσουμε και εμείς την προθεσμία για τις τροπολογίες. Και η συντάκτρια, η συγγήτρια με ενημέρωσε ότι οι τροπολογίες μπορεί να δεχτεί έως την 30 Αυγούστου αύριο δηλαδή στις 12 το μεσημέρι. Ας δώσουμε το λόγο, ας δώσουμε το λόγο στην εισηγήστρια για να μας, εισηγήστρια για να μας εξηγήσει, εξηγήσει. Πολύ κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργία θέλει, θέλει όντως να, όντως να ε, ε, η πρόταση αυτή προκύπτει από το, γεγονός, ότι εντός, τη διατροφική εντός της, ε, ε, διατροφικής, αλυσίδας, παράδειγμα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, η μεγάλες ε, πολυεθνικές του αγροδιατροφικού τομέα και πολύ αδύναμη κρίκη της αλυσίδης, όπως για παράδειγμα η γεωργή. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη συνένεση σε όλες τις χώρες ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν να υπάρξουν αθέμητες ε, πρακτικές, οι οποίες με αυτές τις ε, ανισότητες που υπάρχουν στην εξουσία σίγουρα προκύπτουν. Η κοινή γεωργική πολιτική ήδη έχει εισάγει κάποιες νέες ε, διατάξεις για να βελτιώσει τη θέση στην αγορά, αλλά ακόμα υπάρχει περιθώριο νομοθετικής ευελιξίας. Υπάρχει ένα μέσο το οποίο υπάρχει ήδη που είναι το μέσο της ε, διατροφικής αλυσίδας που είναι ένα προαιρετικό μέτρο και περιλαμβάνει μια σειρά από αρχές καλών πρακτικών που δυστυχώς όμως ε, είναι απόλυτα ανεπαρκές για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες πρακτικές οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης 20 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων η χώρα μου που περιλαμβάνουν εθνική νομοθεσία για τι ε, καταχρηστικές και αθέμητε πρακτικέ όλη τη διατροφική αλυσίδα. και επομένω πιστεύω ότι είναι απαραίτητο και θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το παρουσίασε να υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι κανόνε, ε, ώστε σε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχει προστασία και καταπολέμηση αυτών των πρακτικών. Η πρόταση είναι καλή, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί σε κάποιες πτυχές ώστε να αποφύγουμε να γίνει μία απλή πολιτική δήλωση. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Θα ε, προτείνω κάποιες αλλαγές. Να πω ότι η έκθεση του Πάλο Ντεκάστρο είναι πολύ καλή ε, από την Επιτροπή Γεωργίας που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Καταρχάς, το πεδίο εφαρμογή είναι πολύ περιοριστικό, διότι περιορίζεται μόνο στη σχέση μεταξύ μιας ε, μικρομεσαίας επιχείρησης πολιτή και μιας μικρομεσαίας επιχείρησης αγοραστή και όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την οικονομική στη θέση και στη θέση του στη διατροφική αλυσίδα πρέπει να την χάνουν προστασίας. Προτείνω λοιπόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή και εδώ έχουμε τις τροπολογίες 1, 2, 4, 5 και 8. Επίσης, να πω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν πιο περιοριστική νομοθεσία από αυτή που προτείνει η οδηγία και αυτό το μέτρο πρέπει να ισχύει για όλο το κείμενο και όχι μόνο για κάποια άρθρα όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ έχουμε την τροπολογία 29. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης δεν αναφέρεται ε, στην ε, πώληση με ζημία, που είναι μία από τις πρακτικές που καταγγέλλεται περισσότερο, διότι υπάρχουν ε, προμηθευτές οι οποίοι έχουν ελάχιστο περιθώριο ευελιξίας για να δράσουν λόγω της αβεβαιότητας και των νομικών κενών που υπάρχουν. Και εδώ έχουμε την τροπολογία 17. Στη συνέχεια, οι γραπτές ε, συμβάσεις δεν είναι μόνο ικανή και αναγκαία στη συνθήκη, αλλά είναι αυτό το οποίο συστήνεται για να αποφύγουμε καταχρηστικές πρακτικές οι οποίες οφείλονται στις εγγυήσει που ε, προτείνει ο προμηθευτής. Ε, και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές συμβάσεις σε κάθε κράτος μέλος, αλλά να μπορεί και κάποιος να ε, προσφύγει στα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν ε, να προσβάλλουν αυτές τις συμβάσει και να τις επιβάλλουν ε, στην χώρα τους. Επίσης, δεν υπάρχει, η, υπάρχει μεν υποχρεωτική δυνατότητα συμβάσεων, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυτό το δικαίωμα. Αυτά είναι η τροπολογία 22 με την οποία προσπαθώ να βελτιώσω τη διατύπωση. Ε, θα την ε, ε υποβάλω και τη σχετική τροπολογία αύριο πριν από τις 12. Επίσης, τα, οι γραπτές συμβάσεις για να αποφύγουμε θέμητες πρακτικές πρέπει να έχουν και ένα ενιαίο ε, κριτήριο για να υπολογίζονται κυρώσεις για το θέμα αυτό. Εγώ πρότεινα κάτι αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στην νομοθεσία σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στην Αλία. Ε, και έχουμε την τροπολογία 27 σχετικά, αλλά θα μπορούσε να συζητηθεί και είναι και κάτι το οποίο είναι προσυζήτηση, το αντιλαμβάνομαι, διότι ε, πήρα απλώ κάτι που υπάρχει σε άλλη νομοθεσία. Εάν ε, όμως ε, δεν υπάρχει αυτό, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας για τις κυρώσεις. Και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες εθνικές διατάξεις που ήδη εφαρμόζονται, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, ε, να έχουν εθνικά παρατηρητήρια για τα διατροφικά θέματα για να παρακολουθούν τις τιμές και τις καταχρηστικές πρακτικές. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ε, επιτρέψει και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό στην τροπολογία 28 και αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία έχω να προτείνω εγώ στο σχέδιο γνωμοδότησης και να σας υπενθυμίσω όπως ε, είπατε και εσείς είναι πολύ μικρή η προθεσμία, είναι αύριο το πρωί η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Τελασέσκο. Mulțumesc, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που κατέβαλε να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν. Οι αθέμητες πρακτικές οδηγούν σε σπατάλη τροφίμων και σε μείωση των ποιοτικών προτύπων. Γι' αυτό και πρέπει να μειωθούν οι ανθέμητες πρακτικές στο μέτρο του δυνατού. Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σχετική νομοθεσία. Γι' αυτό και ε, επανέρχεται η Κομισιόν με νέα πρόταση. Όμως δυστυχώς αυτή τη φορά είμαστε, είμαι κάπως απογοητευμένος. Περίμενα η πρότασή της να είναι πιο ολοκληρωμένη και πιο φιλόδοξη. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μια καλή βάση συζήτησης από την οποία μπορούμε ως αφετηρία να ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις μας προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα θετικό κείμενο. Θεωρώ ότι πρέπει καταρχάς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Επίσης, θα πρέπει στον κατάλογο των αθέμητων πρακτικών να προσθέσουμε μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν συγκαταλέγονται σε αυτές τις αθεμητές πρακτικές ώστε ο κανονισμός να ε, περιλαμβάνει έναν εξαντλητικό κατάλογο αθέμητων πρακτικών. Επίσης, η αρχή της μη αποκάλυψης θα πρέπει να εφαρμόζεται, να ε, μην ε, διαγραφεί από τον ε, κατάλογο των κριτηρίων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Γιούσο για την ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σπατάλη τροφίμων, η εκμετάλλευση των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ε, παράγουν τρόφιμα. Υπάρχει και ένα ε, παράδειγμα από την Πολωνία όπου ένα συγκεκριμένο είδος μούρων ε, αγοράστηκε από γεωργούς στα 10 cent και η τιμή πώληση στον τελικό καταναλωτή ήταν πάνω από 4 ευρώ. 40%, 40 ε, φορές πάνω δηλαδή. Πρέπει προφανώς και να ρυθμιστεί το θέμα αυτό ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι θα προτιμούσα το ζήτημα αυτό να ρυθμιστεί σε εθνικό επίπεδο. Επειδή όμως μιλούμε για μεγάλους λιανεμπόρους και χονδρεμπόρους είναι αναγκαίο να υπάρξει ευρωπαϊκή ρύθμιση προκειμένου να περιοριστούν οι πρακτικές αυτές. Συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων βεβαίω, γιατί αν δεν υπάρχει ηθική και δεοντολογία, δυστυχώ το μόνο που μα απομένει είναι η εφαρμογή του νόμου. Και θέλω να, ρωτήσω την ε, εισηγήτρια, για ποιο λόγο ε, έχουν εξαιρεθεί οι συνεταιρισμοί από, από το πεδίο εφαρμογή. Γιατί οι αθέμετες πρακτικέ μπορεί να πλήξουν όλους τους ε, ε, στην αγορά. Θα υποβάλω και εγώ τις τροπολογίες που θέλω έως αύριο το μεσημέρι. Yes, thank you very much, Chair, would like to uh, thank the... Ο κύριος Κουίταμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό ε, έργο. Προφανώ όλοι διαφωνούμε με τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ και συμφωνούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό και με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το στόχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε λοιπόν μια μελέτη αντικτύπου, ε, αντικτύπου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προστατευτούν οι πλέον αδύναμοι, εκείνοι που έχουν τη μικρότερη διαπραγματευτική δύναμη στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια δίκαιη και σαφής αλυσίδα εφοδισμού τροφίμων η οποία θα δίνει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους. Αυτό που βλέπω τώρα να προσπαθούν οι συνάδελφοι να κάνουν με τις τροπολογίες είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και στην ομάδα μου είναι να διευρυνθεί η πρόταση, το πεδίο εφαρμογής της πρότασης κομισιών Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να επιλύουμε προβλήματα τα οποία, προβλήματα τα οποία δεν υπάρχουν ούτε χρειάζεται να Βεβαίω και πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και αρνητικέ επιπτώσει αν διευρυνθεί υπερβολικά το πεδίο εφαρμογή. Ενδεχομένω, ε, να υπάρχουν και κάποια θετικά επιχειρήματα υπέρ μια τέτοια κίνηση. Ε, οπότε αυτό που μου απομένει να κάνω είναι για ποιο λόγο, να ρωτήσω την Κομισιόν για ποιο λόγο επέλεξε το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή που προτείνει και τι ε, θεωρεί εκείνη, τι πιστεύει εκείνη ε, σχετικά με τι προτάσει διεύρυνση αυτού του πεδίου εφαρμογή. Δεύτερον, υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών στη στάση τους. Κάποια κράτη-μέλη ε, διαθέτουν εθνική νομοθεσία η οποία αντιμετωπίζει και καταπολεμά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές άλλα κράτη-μέλη έχουν λιγότερο τελειοποιημένη ε, εθνική νομοθεσία να το πω έτσι. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα θετικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, να υπάρχει και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο πεδίο η εθνική νομοθεσία προκειμένου να αντιμετωπιστούν ε, τέτοιου είδους πρακτικές. Δεν μπορεί να θεωρούμε, δεν, δεν θεωρώ, εν πάση ε, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να θεσπίσουμε νομοθετικά μια πανάκια εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, είμαι ανοιχτό στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κονέτσνα. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, είναι ε, βεβαίως είναι σημαντικό αυτό το θέμα που έχει επιπτώσεις πάνω σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τη συζήτηση, λυπούμε, διότι αυτή η γνωμοδότηση θα έχει αντίκτυπο ζωτικό για τους γεωργούς, για τους πολίτες, για την ύποθρο, διότι υπάρχουν στα κράτη-μέλη ορισμένες, ορισμένοι κανόνες που είναι κατακαιρματισμένοι. Ε, είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και είναι ασυμβίβαστες. Οι μηχανισμοί συντονισμού μας λείπουν τα σημεία που με ανησυχούν σε αυτή τη γνωμοδότηση πρέπει να συζητηθούν, προετοιμαστούν καλύτερα ότι έχουν συνέπειες πάνω στα κράτη-μέλη. Όταν μιλάμε για τις σχέσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε ε, υπάρχουν ε, αθέμητοι ε, αθέμητες πρακτικές που δεν τις αφορούν μόνο. Υπάρχουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ε, τροφίμων αυτές οι αθέμητες ε, πρακτικές. Δεν έχουμε τον ορισμό των αθέμητων πρακτικών. Τι είναι ακριβώς μια, ένας αθέμητος ε, ανταγωνισμός. Υπάρχει ένας κατάλογος σε διάφορα κράτη-μέλη οι επιχειρήσεις έχουν μάθει πώς να παρακάμπτουν ε, τους κανόνες αυτούς περί αθέμη του ανταγωνισμού. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν πάνω από 30 ε, θέμητες ε, πρακτικές. Εξαφανίζεται μια πρακτική, εμφανίζονται δύο. Έχουμε πολυεθνικές εταιρείε αγροτροφικές που συμφέρονται κακώς στα κράτη-μέλη και η Κομισιό δήθεν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι κανόνες είναι ανεπαρκείς, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις συμβάσεις που έχουν συναυθεί. Αλλά όλες οι σχέσεις δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις. Αν είναι οι συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, ε, δεν είναι μόνο οι συμβάσεις, πρέπει να περιλαμβάνονται και οι σχέσεις μεταξύ πολιτών και αγοραστών. Υπάρχουν ε, διάφορα λάθη ε, στην γνωμοδότηση και δεν βοηθούν τους μικρούς, διότι αυτή η οδηγία υποστηρίζει τα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη δηλαδή δίνει την δυνατότητα στις πολυεθνικές να δράσουν με βάση το χρήμα οι μεγάλες πολυεθνικές. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αναπέμψουμε στην Κομισιόν το θέμα αυτό. Αλλά εφόσον δεν έχουμε χρόνο, ετοίμασα 105 τροπολογίες και θα αγωνιστώ ε, για να υιοθετηθούν. Ευχαριστώ. Με μόνο την αγγλική εκδοχή. Ο κύριο Λαβία. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που έκανε διότι σε 20 από τις 27 παρούσες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση ήδη υπάρχει εθνική νομοθεσία, αλλά δυστυχώ δεν λειτουργεί σε πολλές χώρες και επομένω, επειδή ε, έχουμε και διεύρυνση των εμπορικών ανταλλαγών, χρειαζόμαστε κοινού κανόνε. χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση με την οποία φυσικά είμαι απόλυτα υπέρ. Συμφωνώ πολύ με τα όσα έκανε η συντάκτρια για πρόταση διεύρυνση, όχι μόνο για τα διατροφικά προϊόντα, αλλά για όλα τα γεωργικά προϊόντα, ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και κάποιε άλλε μορφέ ε, προϊόντων, τα οποία εξαιρούνται από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει επίση να ρυθμίσουμε και κάποιε συγκεκριμένε πτυχέ που αφορούν ε, τι ε, ε, πωλήσει κάτω του κόστου, τι εκπτώσει που γίνονται στο τέλο του όχρη, οι οποίε είναι ει βάρο των πιο αδύναμων κρίκων τη αλυσίδα δηλαδή των ε, παραγωγών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις πρώτες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει το θέμα των συμβάσεων, αλλά οι συμβάσεις είναι τελείως διαφορετικές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει εξομάλωνση των συμβάσεων και να υπάρχουν και κάποιες συνέπειες ε, και θετικός αντίκτυπος όμως, αλλά τουλάχιστον για κάθε χώρα να βοηθάμε ε, και σε κρατικό επίπεδο, όπως έγινε σε κάποιες χώρες και είχαμε με θετικά αποτελέσματα. Επίσης υπάρχει και το θέμα των συμβάσεων μεταξύ ατομικών στοιχείων της αλυσίδας. Αυτό σε κάποιες χώρες λειτουργήσε, σε κάποιες άλλες ε, είχε αρνητικό αντίκτυπο. Επομένως θα πρέπει να γίνει με ενιαίο τρόπο η λύση του θέματος, ώστε να μην μπορεί να το ε, στρεβλώσει κανένας και να αποτελέσει και βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε να έχουμε ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Και ένα τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος, οι συνέπειες αυτής της νομοθεσίας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες θα είναι εις βάρος αυτού που δεν είναι ο αδύναμος κρίκος, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος, ε, κυρίως ένα ε, ακροδιατροφικό σύστημα το οποίο είναι ολένα και πιο κατακαιρματισμένο, να πλήξουμε τους λιγότερους χειρούς, αυτούς που έχουν λιγότερη εμπορική δύναμη, αυτούς που δεν είναι σε θέση να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο όγκο των ε, μεγάλων σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέγκελε τώρα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι, διότι σχεδόν έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η πρόταση είναι αποτέλεσμα μιας ε, μακροσκελούς και μακράς διαδικασίας, η οποία διέρχησε πάνω από 10 χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μας όλα τα στάδια. Τελικά λοιπόν πιστεύω ότι καταφέραμε να έχουμε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα ώστε να ε, προτείνουμε την οδηγία που σας προτείναμε. Βεβαίω, ε, πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να εγκριθεί η οδηγία πριν από το τέλο ε, τη κοινοβουλευτική θητεία. και αυτό είναι αυτό το οποίο ε, συζητήσαμε και με του συναδέλφου σα στην Επιτροπή Γεωργίας και νομίζω ότι ο κύριο Δεκάστρο είναι αναφανδόν υπέρ αυτές τη προσέγγιση. γιατί κανεί δεν ξέρει τι θα απογίνει η πρόταση εάν δεν εγκριθεί εντό τη παρούσα θητεία. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να το εκμεταλλευτούμε. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έθιξε η συντάκτρια τη νομοδότηση και ο κύριο Χούιταμα είναι το θέμα τη επέκταση του πεδίου εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να προστατεύσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει έναντι των μεγάλων ε, λιανοπολιτών διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, προστατεύσουμε του αδυνάμου ε, έναντι των ισχυρών. Και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγο να προστατεύσουμε πολυεθνικές ε, Παραγωγού τροφίμων ε, για ε, έναντι μικρών παραγωγών. Γιατί να προστατεύσουμε την Καρφούρ και τη Unilever εναντίον της Καρφούρ. Δεν έχω δει κάποιο έγκυρο, ισχυρό επιχείρημα που να το εξήγει αυτό. Το δεύτερο επιχείρημα είναι νομικής φύσεως, διότι εδώ είμαστε στο άρθρο 43 της συνθήκης, που είναι η γεωργική νομική βάση πρέπει να φροντίσουμε να μην υπερβούμε τα όρια και να μην απομακρυνθούμε πάρα πολύ από το γεωργό, που είναι αυτός ε, ο οποίος ε, ε, θέλουμε να προστατεύσουμε τελικά. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ δύο μη γεωργικών φορέων, όπως για παράδειγμα μια μεγάλη πολυεθνική παραγωγό τροφίμων και έναν λιανοπολιτή είναι κάτι το επικίνδυνο από νομική σκοπιά και το αναλύσαμε πάρα πολύ προσεκτικά και αυτό είναι ο λόγο που παραμένουμε σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προτείνουμε οδηγία που στόχο έχει να εξασφαλίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελάχιστη εναρμόνιση. Και γιατί ελάχιστη εναρμόνιση, διότι όπω ακούστηκε υπάρχουν ήδη 20 κράτη-μέλη που έχουν νομοθεσία τελείω διαφορετική και επίση 7 κράτη-μέλη που δεν έχουν τίποτα δεν υπάρχει τίποτα από πλευρά νομοθεσία. Ε, Επομένω, ε, η ιδέα είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ενό πεδίου στο οποίο υπάρχει νομοθεσία τελείω διαφορετική μεταξύ τη κάθε χώρα και δεν υπάρχει σημεία χώρες στην οποία δεν υπάρχει καμία νομοθεσία και όλα αυτά να μπορέσουμε να τα συμβιβάσουμε. Και πιστεύουμε ότι με την προσέγγιση τη ελάχιστη εναρμόνιση αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε και γι' αυτό ακριβώ έχουμε ε, εντοπίσει τι πιο ζημιογόνες εμπορικές πρακτικές, ε, τις οποίες ε, αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη, κάποια άλλα όχι και έχουμε ορίσει κατά την άποψή μας με απλό τρόπο. Ε, αυτό συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και με το γεγονός ότι αυτά τα οποία προτείνουμε πρέπει να ασχοληθούν και με την ε, ιδιωτική αυτονομία, που είναι βασική αρχή του ιδιωτικού δικαίου. Να κάνω και μερικά σχόλια για κάποιες τροπολογίες που πρότεινε η συντάκτρια. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τρεις τροπολογίες, τη 18, την 20 και την 21, που αυξάνουν τον αριθμό των πρακτικών. Η διατύπωση αυτών των πρακτικών σε αυτές τις τροπολογίες είναι τόσο ευρεία που πιστεύω ότι τελικά θα οδηγήσουν από την ελάχιστη εναρμόνιση στην πλήρη εναρμόνιση, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει εδώ. Επίσης, θα ήθελα να κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις για κάποιες τροπολογίες, πολύ λίγες, και να σχολιάσω. Ξεκινώ με την τροπολογία 8, που αποκλείει τους συνεταιρισμούς από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Δεν ε, καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ε, παραγωγή που συμμετέχουν σε συνεταιρισμές ε, που τελικά έχουν οδηγήσει σε αρκετά μεγάλους φορείς και τους αρνούμαστε το δικαίωμα να υπερασπίσουν αυτούς ε, για ρήτρε οι οποίες θεωρούμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αυτό δεν συνάδει ούτε με τον αριθμό των διατάξεων στην ΚΑΠ που επίσης ασχολείται και με τις συμβατικές σχέσεις και, με το καταπο... και στο... στις οποίες καλύπτονται και οι συνεταιρισμοί. Επόμενη τροπολογία, η 17, που αφορά τις πωλήσει κάτω του κόστους. Καταρχάς, αυτή είναι μια έννοια που πολύ δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει ανάγκη να δούμε και το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό αυτών των επιχειρήσεων για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να τα εφαρμόσουμε λογικά αυτό. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι πολύ αμφισβητήσιμο και επίση θεωρούμε ότι δεν καλύπτεται το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, διότι δεν είναι μια πρακτική η οποία διαδραματίζει ρόλο στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Το τρίτο είναι για την τροπολογία 22 για τις γραπτές συμβάσεις. Αυτό που προτείνει η τροπολογία είναι κάτι το οποίο μπορούν ήδη τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη ήδη μπορούν να συνάψουν γραπτές συμβάσεις και να είναι υποχρεωτικές αυτές. Δεν χρειάζεται να τους το πούμε εμείς στην οδηγία. Υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις στον κανονισμό ΚΟΑ, ο οποίος επιτρέπει στον πολιτή να ζητήσει γραπτή σύμβαση. Επομένως, ε, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Και κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, η τροπολογία 27 για τις ποινές. Δέχομαι ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια κριτήρια ε, σε κάποια σημεία για να ρυθμίσουμε τις ε, ποινές. Αλλά αυτό το οποίο προτείνει η τροπολογία, να το πω ειλικρινά, είναι δρακόντια μέτρα 2% του κύκλου εργασιών για μία, αυτό αφορά επιχείρηση σαν την Carrefour και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο εξέτασα που έχει κύκλο εργασιών 65 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό θα οδηγήσει σε χρηματική ποινή 1,3 δις ευρώ. Ε, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε αυτό το θέμα. Ε, σίγουρα είναι δυσαρλάλογο και ιδίως ε, όταν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω αύξηση για μη συμμόρφωση και μη σεβασμό ε, συγκεκριμένων εμπορικών πρακτικών. Για να ολοκληρώσω λοιπόν κάνω έκκληση ε, για να έχουμε την προσέγγιση που έχουμε προτείνει εμείς, την ελάχιστη εναρμόνιση που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα ενταχθεί με αρμονία στο ε, ένωμη τάξη των κρατών μελών και θα επιτρέψει να καταλήξουν σε συμφωνία τα θεσμικά όργανα εγκαίρως πριν το τέλος της ε, θητείας του Κοινοβουλίου, χωρίς ε, να υπερφορτώσουμε το καράβι με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κυρία Γιούζο, μόνο αγγλικά από εδώ και πέρα. Θα σταματήσει η διερμηνία. Voy a tratar de ser, eh, muchas gracias a todos